Καλημέρα σας. Δεν είμαστε και τόσοι πολλοί, αλλά έχουμε καθυστερήσει, έτσι. Ναι. Πολλές αλλαγές σημειώθηκαν στην ημερήσια διάταξη, επειδή συνάδελφοι μα είπαν ότι αδυνατούν σήμερα, αλλά και άλλοι που έχουν προσυπογράψει. Εδώ έχουμε την ετήσια έκθεση με τον συνάδελφο Μακμίλαν Σκοτ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επίση αναφορέ που έχουν να κάνουν με τα διορθωτικά ταμεία και τα ε, θέματα ατόμων με άτομα, με, με πρόβλημα για αεροδρόμιο, ότι θέματα ιδιοκτησία στην Κύπρο, επίσης θέματα στην Ουγγαρία και για τα ζώα, διάφορα πειράματα, στα καλλιντικά. Έχουμε αρκετέ μεταβολέ πάντω στην ημερήσια διάταξη για ανάγκες διάφορες, εντάξει, συμφωνώ με τους συντονιστέ. συμφωνήθηκα μόνο αυτές με τους συντονιστές χθες και είπαμε ότι πραγματικά χρειαζόταν να αλλάξουμε και την ώρα έναρξης αλλά και εξέτασης και τις διάφορες αλλαγές. Σας γνωστοποιήσαμε αυτές τις αλλαγές και να σας πω ότι το σημείο 5, δηλαδή την έκθεση ετικά με τη διερευνητική επίσκεψη στη Γαλλική, αυτή αναβλήθηκε την επόμενη φορά γιατί το δεν συντάχθηκε πλήρως από τα μέλη της Επιτροπής το σχετικό κείμενο και αναβάλαμε την εξέταση του σημείου αυτού. Και επίσης η οδηγία για τις κλιματικές επιπτώσεις με τον κύριο Χουντή θα εξεταστεί, μας το ζήτησε ο ίδιος ο κύριος Χουντής στις 3 το απόγευμα. Θα ξεκινήσουμε με το σημείο 13, δηλαδή με εγκατάσταση δύο ελικών πάρκων στη μεθαρική περιοχή της Τσεχίας ε, και της ε, επιβλαβείς επιπτώσεις στη Γερμανία. Και εδώ τα υπόλοιπα είπαμε έχουν αναβληθεί. Θα το εξετάσουμε αυτό πρώτο και επίσης για τα ε, δικαιώματα για τα θετικά ταμεία και για τα προβλήματα ατόμων ε, θα εξεταστούν αργότερα σήμερα και μετά θα έχουμε και τα σημεία 9 και 10 με το ίδιο θέμα πάντα και ο συνάδελφος Μακμίλαν Σκοτ θα κάνει τις πρώτες εκτιμήσεις του για την ετήσια έκθεση της Επιτροπής Αναφορών στις 11 παρατέταρτο περίπου, πριν από τη συνάντηση δηλαδή των συντονιστών. Και σήμερα το απόγευμα θα επαναλάβουμε τις εργασίες μας, θα πούμε τι αποφάσισαν οι συντονιστές και μετά με την έκθεση του κυρίου Χουντή, όπως είπαμε. Θα ασχοληθούμε και με διάφορες αναφορές για την εγκατάσταση, ας πούμε, αεροδρομίου στην Notre Dame de και οι αναφέροντες αρκετοί θα είναι παρόντες και ακούσαμε ότι θα παραστούν και υπογράφοντες ε, την ε, αναφορές του 8, 9, 10, 15, 17 και 18. Δεν έχω κάτι να συμπληρώσω. Και παρακαλώ συνάδελφοι, μήπως θέλετε εσείς ε, εγκρίνετε ακριβώς τη σημερινή για διάταξη με τη μορφή αυτή. Κυρία Τζανόσκα. Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Μπορείτε να επαναλάβετε παρακαλώ. Από αυτά που έχουμε τώρα, μπορείτε να μας τα εξηγήσετε σιγά σιγά ποια θέματα θα εξετάσουμε σήμερα, ποιες ερωτήσεις, δε, ποιες αναφορές θα εξετάσουμε σήμερα, γιατί δεν σας κατάλαβα με τη σειρά. Λοιπόν, να τα ξαναπούμε. Άλλαξε η μερίσια διάταξη από το Προεδρείο. Να σας πω ότι θα ξεκινήσουμε με την αναφορά στο σημείο 13. Αυτό θα είναι το πρώτο θέμα μας. Εντάξει, να σας το πω και αγγλικά, το 13. Στη συνέχεια, περνάμε στα σημεία 8, 9 και 10. Μετά, έχουμε τη γνωμοδότηση Μακμίλαν Σκοτ, που είναι το σημείο 7. Μετέχουμε έχουμε συντονιστές, αυτά για το πρωί. Και το απόγευμα αρχίζουμε με τον κύριο Χουντή, το σημείο 6 δηλαδή. Και μετά το 14. Συμφωνείτε? Καλώς. Δεύτερο σημείο, έγκριση πρακτικών της συνάντησης του Ιανουαρίου και των προηγούμενων συνεδριάσεων ακριβώς. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει μια κάποια παρατήρηση, τότε εγκρίνονται τα πρακτικά. Για το σημείο 3 τώρα, να ανακοινώσω κάτι κάτι που ζήτησε από πλευρά Μάγερ να παραμείνουν ε, ανοιχτές οι 1408 του 2010 και 1157 του 2010 επίσης για εξορυκτικές ε, δραστηριότητες στη Μορόβια. Τελευταία ανακοίνωση για τους συναδέλφους και για τους υπαλλήλους της Επιτροπής. Μας είπε κ. Μποζούτιλ ε, να εγκαταλείψει, να παραιτηθεί από εδώ γιατί έχει εκλεγεί στο Κοινοβούλιο της Μάλτας και θα θέλαμε στο συνάδελφο να τον χαιρετήσουμε και να τον ευχαριστήσουμε για τη συνεργασία μας αυτά τα τελευταία χρόνια με μας όλους αλλά και με τη γραμματεία όπως επίσης ε, και εκ μέρου των Ευρωπαίων πολιτών και εξ ονόμα της Επιτροπής μας του απευθύνω ευχές για πολύ καλή και σωστή δουλειά. Πάμε παρακάτω τώρα, ξεκινάμε με την ημερήσια διάταξη τη νέα την τροποποιημένη. Ξεκινάμε με την 1160 του 2009 του Βέρνερ Σάντιγκ. Απόνομος ο αναφέρον. Γι' αυτό το λόγο έχει από πλευράς Επιτροπής ε, Γκουτμαρ Κόπμαν. Καλή σας μέρα κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί τις εξελίξεις από το 2009, τότε δηλαδή που έφτασε η αναφορά. Έχουμε να κάνουμε εδώ με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και με την εφαρμογή του άρθρου 4 της οδηγίας IA ε ε και με την οδηγία επίσης για τους οικότοπους. Το σχέδιο λοιπόν αυτή τη στιγμή περνάει από την διαδικασία του IA. Ε Δεν έχει δοθεί η άδεια ακόμα και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί αυτό το μήνα. Έχουμε πάρει συγκεκριμένες ερωτήσεις βέβαια από τον κύριο Γιάρ, γι' αυτό και θα ήθελα να δώσω απαντήσεις. Η πρώτη ερώτηση έχει να κάνει με την αξιολόγηση που έγινε από γερμανική και τσεχική πλευρά. Οι τσεχικέ αρχές όμω πρέπει να αξιολογήσουν το πρόγραμμα. Κοινοποιήθηκε στις γερμανικές αρχές το πρόγραμμα βάσει του άρθρου 17 της οδηγίας. Επίσης υπήρξε και διαβούλευση με το κοινό, όπως απαιτείται από το άρθρο 7α τη ε, ίδια οδηγία. Δεύτερη ερώτηση. Έχει να κάνει με δεχόμενη προσφυγή. Η Επιτροπή εξέτασε ε, την υπόθεση βάσει της αρμόδιας υπηρεσίας της Τσεχίας και ε, δεν υπάρχουν ενδείξεις για προβλήματα. Τρίτη ερώτηση. Έχει να κάνει με την παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν ενήμερη για κάποια προσφυγή. Όχι, γιατί δεν υπήρξε προσφυγή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τώρα. Η τελευταία ερώτηση ήταν κατά πόσο χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκά κονδύλια το πρόγραμμα ή όχι. Εφόσον δεν υπάρχει άδεια ακόμα και δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, προφανώς και δεν στηρίζεται με ευρωπαϊκά κονδύλια. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που ε, μπορούσαμε να βάλουμε το θέμα αυτό στο αρχή της ημερήσιας διάδοξης. Η Κομισιόν ε, απάντησε επισήμως, αλλά το πρόβλημα είναι ότι εδώ μιλούμε για ένα project όπου οι επιπτώσεις του είναι διασυνοριακές, γιατί μιλούμε για τα σύνορα μεταξύ Γερμανίας και Τσεχικής Δημοκρατίας. Εκεί θα γίνει το ε, αιωλικό πάρκο με 35 έως 70 μέτρα ανεμογεννήτριες, σε γυπνίαση δηλαδή, ε, και μιλούμε και για μια ε, περιοχή που είναι προστατευόμενη. Οπότε τα, οι ε, συνέπειε του αεολικού πάρκου θα πρέπει να μελετηθούν όχι μόνο για την ε, τσεχική πλευρά αλλά και για την ε, γερμανική πλευρά και σε διαφορά αφορά το περιβάλλον κτλ. Μιλούμε για γυτνία σε 35 έως 70 μέτρων. Ε, προφανώς αυτό θα, θα επηρεάσει και την γενική κατάσταση στην περιοχή Εμεί θεωρούσαμε ότι εκεί θα μπορούσε η περιοχή να αναπτυχθεί και σε ό,τι αφορά την ομορφιά τη περιοχή και τον τουρισμό που έρχεται για την ε, ομορφιά τη περιοχή. Οπότε υπάρχουν κάποιε αμφιβολίε ακόμα για το κατά πόσο θα παραμείνει προστατευόμενη περιοχή η περιοχή αυτή που θα γίνει το νέο ολικό πάρκο. Το πρόβλημα για μένα έχει να κάνει το είπε σωστά η Κομισιόν, ότι βεβαίως υπάρχει όλη η διαδικασία που εξελίσσεται, έχουν ξεκαθαριστεί οι όροι του παιχνιδιού, τα θα, το υλικό πάρκο αυτό θα εγκατασταθεί στην τσεχική πλευρά. Ε, υπεύθυνη λοιπόν για την διεξαγωγή όλων αυτών θα είναι η τσεχική πλευρά, αλλά βεβαίως εδώ υπάρχει μια αντίφαση ότι η αξιολόγηση των τσεχικών αρχών είναι τελείως αντίθετη με την αξιολόγηση των ε, γερμανικών αρχών. Εδώ δεν μιλούμε λοιπόν για θέμα πεποίθησης, δεν μιλούμε για θέμα θεωρητικό, για θέμα αξιών, αλλά μιλούμε για το ότι υπάρχουν αντίθετα τελείως στοιχεία για, ανάμεσα στις δύο αξιολογήσεις των δύο χωρών. Οπότε τώρα το ερώτημα είναι οι ίδιες ευρωπαϊκές οδηγίες, οι ίδιες απαιτήσει, τα ίδια καθήκοντα που έχουν τα κρατη πώς είναι δυνατόν να οδηγούν αυτά τα ίδια κείμενα σε τόσο διαφορετικά αποτελέσματα. Ε, και βεβαίως η Κομισιόν λέει τι θα κάνουμε σε μια τέτοια περίπτωση. Έχουμε ένα, μια περιοχή η μία περιοχή έχει την ιδιοκτησία γιατί εκεί θα γίνουν οι εγκαταστάσεις και τι γίνεται όπου τα δύο κράτη-μέλη έχουν τελείως διαφορετική αξιολόγηση της κατάσταση. Και οι δύο έχουν γνωμοδοτήσεις και οι δύο έχουν κάνει τις αξιολογήσεις τους, τις αναλύσεις τους, οπότε ρωτώ την Κομισιόν. Ε, ασχολούμαστε στην Επιτροπή με την ε, εξέταση της ε, περιβαλλοντικής ε, ε, ανθεκτικότητας. Πρέπει να υπάρξει κάποιο, κάποιο όριο, κάποιο ανόφλη. Νομίζω λοιπόν ότι η τσεχική πλευρά κινείται πολιτικά κυρίως για να χτίσει αυτό το αιωλικό πάρκο. Ερώτημα λοιπόν, τι γίνεται όταν δύο κράτη-μέλη για το ίδιο πράγμα καταλήγουν σε δύο τελείως διαφορετικές, για να μην πω αντικρουόμενες αναλύσεις. Η δεύτερη ερώτηση. Και για τα αιωλικά πάρκα βέβαια, αυτό είναι αρκετά δύσκολο. Όταν εγκριθεί αυτό το project, και μετά ξεκινήσει η διαδικασία. Και ε, αναδρομικά φτάσουμε στο αποτέλεσμα ότι έχουν υπάρξει λανθασμένοι υπολογισμοί. Δεν πρέπει να γίνει κάτι. Δεν πρέπει ας πούμε να κλείσει το, α, το αιωλικό πάρκο μετά, ε, μετά από 6 μήνες. Ναι, αλλά μέχρι τότε θα έχουν χτιστεί κάποιες εγκαταστάσεις. Ε, τι θα γίνει. Το ερώτημα λοιπόν για τέτοια project, ακριβώς που, επειδή έχουν και πολύ σύντομο διάστημα για την, ε, ε, για την ε, διεξαγωγή τους, είναι πώς μπορούμε θεωρη, να αξιολογήσουμε τα πράγματα τόσο εις βάθος, για να μπορέσουμε να μην καταλήξουμε τελικά σε λαθασμένα συμπεράσματα, σε λαθασμένα αποτελέσματα που θα πρέπει μετά αναδρομικά να τα διορθώσουμε. Γιατί όλα αυτά βεβαίως κοστίζουν χρήματα, έτσι. Δεύτερο ερώτημα λοιπόν. Η Κομισιόν πώς μπορεί να είναι σίγουροι ότι θα γίνει αυτή η βάθος ανάλυση για να μην υπάρχουν μετά αρνητικές συνέπειες και ανάκληση των σχεδίων. Και ένα τρίτο ερώτημα που έχω, η Κομισιόν πώς αξιολογεί και ποιες είναι οι δυνατότητες που έχει για τις ε, πρωτοβουλίες των πολιτών. Γιατί μιλούμε για κρατικές αρχές οι οποίες επεμπλέκονται βεβαίως, Πάλι λέω ότι είναι διαφορετικέ οι αναλύσει των δύο χωρών από αυτού. Τρίτο ερώτημα λοιπόν, οι, οι πρωτοβουλίε των πολιτών τι μπορούν να, πώς μπορούν να βοηθήσουν σε ό,τι αφορά και την εποπτεία ίσω. Τι μπορούν να κάνουν όταν, είναι την, όταν έχουν την άποψη ότι η αξιολόγηση των ε, επίσημων αρχών είναι τελείως αντίθετη σε αυτά που πιστεύουν. Ένα τέταρτο ερώτημα που είχα το απάντησε η Κομισιόν, οπότε το σημειώνω, σημειώνω την απάντησή της, ότι η Τσεχία δηλαδή για την ε, δημιουργία αυτού του υλικού πάρκου δεν έχει λάβει οικονομική ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Επιτροπή λοιπόν πρέπει να ασχοληθούμε πολύ εντατικά με το θέμα αυτό. Τι κάνουμε με αυτές τις αξιολογήσεις ε, για το περιβάλλον ε, ε, και πώς μπορούμε να διχειριστούμε δύο τελείως διαφορετικές αντικρουόμενες αναλύσεις αξιολογήσεις από τα κράτη-μέλη. Γιατί όταν το ένα κράτος μέλος ε, έχει όλη την ευθύνη, προφανώς το άλλο κράτος μέλος ε, ε, έχει νιώθει ότι υποβιβάζεται σε αξία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον ομιλητή. Ο εκπρόσωπο της Επιτροπής, κ. Χόφμαν, θα μπορούσε να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα που ακούστηκαν. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Όπως είπα και πριν, Εξαρτάται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία το σχέδιο αυτό. Υπάρχει η αδηγία, υπάρχει σύμβαση, σύμφωνα με τα οποία οι τσεχικές αρχές πρέπει να αξιολογήσουν το πρόγραμμα. Οι, γενικές, οι γερμανικές αρχές έλαβαν κοινοποίηση σχετικά με το πρόγραμμα αυτό και το γερμανικό κοινό έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στη διαδικασία. Ενημερωθήκαμε για το ότι το κοινό στη Γερμανία συμμετείχε στη διαδικασία συμμετείχαν στην ε, δημόσια συζήτηση η οποία οργανώθηκε τον Φεβρουάριο που μας πέρασε και εκεί έγιναν και τα διάφορα ζητήματα που τους απασχολούν. Εάν υπάρξει προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εννοείται ότι θα εξετάσει αδελεχέστερα την υπόθεση. Δεν υπάρχει όμως προς το παρόν τέτοια προσφυγή. Η αξιολόγηση που έκανε η Γερμανία δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη γιατί δεν συνάδει με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Αυτά όσον αφορά την πρώτη ερώτηση. Έρχομαι τώρα ε, στο κατά πόσο μπορεί να κλείσει το πρόγραμμα. Δεν έχει υπάρξει αδειοδότηση για το πρόγραμμα προς το παρόν. Συνεπώς δεν υφίσταται το πρόγραμμα αυτό, το σχέδιο αυτό. Και παρόλο που αναμένουμε οι τσεχικές αρχές να ε, καταλήξουν στο κατά πόσο θα έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις ή όχι το σχέδιο αυτό, προς το παρόν δεν υπάρχει καμία παραβίαση του κοινοτικού δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν βρίσκει καμία τέτοια παραβίαση. Στα τέλη αυτού του μήνα, από ό,τι φαίνεται, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία και οι τσεχικές αρχές θα έχουν καταλήξει για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον τόσο από πλευρά Τσεχίας όσο και Γερμανίας και βάσει των συμπερασμάτων αυτών τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίσως να μπορέσει να δράσει εφόσον κάτι δεν πάει καλά. Όσον αφορά τώρα τις κινητοποίησεις των πολιτών, ε, βεβαίως και θέλουμε την ε, αντίδραση των πολιτών, αλλά βλέπετε ότι τα δικαιώματά τους στηρούνται πλήρως. Η επιχειρηματολογία που χρειάζεται έχει προσφερθεί και στα γερμανικά από τις τσεχικές αρχές. Οι τσεχικές αρχές κοινοποίησαν ε, και ενημέρωσαν την Γερμανία για το πότε γίνεται διαβούλευση με το κοινό και έτσι οι πολίτες από πλευράς Γερμανίας είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στη διαβούλευση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την Κομισιόν που μου απαντά. Έχει δίκιο. Η απόφαση δεν έχει ληφθεί ακόμη. Το είπε και η Κομισιόν μέχρι το, μέχρι το τέλος του μηνός την περιμένουμε. Οπότε μόνο τότε μπορούμε να προσφύγουμε εφόσον έχει ληφθεί η απόφαση η δική μου παράκληση είναι ότι μόλις ληφθεί η απόφαση και, μάλλον, και όλα μάλλον δείχνουν ότι θα υπάρξει μια πολιτική απόφαση από την τσεχική κυβέρνηση να εξετάσουμε γρήγορα το τι γίνεται γιατί ε, σας είπα ότι είναι πολύ λίγος ο χρόνος με το, από την απόφαση και μετά μέχρι να γίνει το πάρκο Οπότε αυτό ήταν το δικό μου το αίτημα, να κάνουμε μια σωστή ενδελεχή εξέταση. Αυτή τη στιγμή ληφθεί η απόφαση για να δούμε κατά πόσο μπορούμε μετά να προσφύγουμε κτλ. Το δεύτερο που πρέπει να πω είναι ότι από, την, από τη μία έχουμε πραγματικά μεγάλο άχθος, αποκινούμε τα κράτη-μέλη, έχουμε ορίσει τους ε, προστατευό, τις προστατευόμενες περιοχές, αυτό ήταν καλό και Απ' τη μία έχουμε ε, ορίσει αυτές τις προστατευόμενες περιοχές. Ε, προφανώς ε, κάποιες ε, πρακτικές για την εγκατάσταση τέτοιων υλικών πάρκων δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή δεν θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Γιατί αλλιώ τι να τα κάνουμε, τι να τι κάνουμε τι προστατευόμενες περιοχές; όταν μπορούμε να χτίσουμε παντού. Θα πρέπει λοιπόν κάποιες πρακτικές, κάποιες τέτοιε διαδικασίε να να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για να, προστατευτεί και ο, να προστατευτούν και οι πολίτες από τις δύο πλευρές των συνόρων. Τώρα, η επικοινωνία μεταξύ των δύο χωρών ε, ε θα μπορούσε να βελτιωθεί προφανώ. Είναι άλλη ιστορία όμω αυτή. Θα μπορούσαμε να το προσπαθήσουμε. η Κομισιόν είπε ότι έχει γίνει όλη η διαδικασία διαβούλευση, αλλά και πάλι λέω ότι όλα αυτά θα γίνουν και μετά την λήψη τη απόφαση. Οπότε α την αφήσουμε την υπόθεση αυτή ανοιχτή μέχρι να ληφθεί η απόφαση. Και μετά να επανέλθουμε και να ξανασυζητήσουμε. Και ζητώ πάλι από την Κομισιόν, αυτή τη στιγμή ληφθεί η απόφαση, όπω περιμένω ότι θα γίνει, υπέρ δηλαδή τη εγκατάσταση του ελληνικού πάρκου, η Κομισιόν σύντομα, άμεσα, να εξετάσει τι προσφυγέ που υπάρχουν κατά αυτή τη απόφαση και να δει κατά πόσο όλα αυτά έχουν γίνει με, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Ευχαριστώ. Παραμένει ανοιχτό το θέμα λοιπόν γιατί προβαίνει σε παληθεύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με όσα ζητήσουν οι αναφερόμενοι και όπω ο σνάθο Γιάρ ζήτησε περιμένουμε να μα ενημερώσει η Επιτροπή για το πώ εξελίσσεται η κατάσταση. και μετά από ένα κάποιο χρονικό διάστημα θα ζητήσουμε τις απαντήσεις ε, εξ ονόματος ακριβώς των πολιτών που τις ε, ζητούν. Κλείνουμε το σημείο αυτό της ημερήσιας διάταξης, να πάμε στο επόμενο σημείο. Είναι το σημείο 8 η αναφορά της Τζούντιθ Κλάιν, η θα ηθαγένειας, παρούσα η αναφέρουσα και έχει το λόγο ακριβώς για να μας πει πώς έχει το θέμα το οποίο θέτει με την αναφορά της. Πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Η αναφορά μας έχει να κάνει με την κατάχρηση που γίνεται στα διαρθρωτικά ταμεία από ορισμένε χώρε μέλη, οι οποίε κάνουν διακρίσει σε βάρο των ατόμων με αναπηρίε. Και γιατί, γιατί οι εκατοντάδε χιλιάδε ευρώ δεν επενδύονται σε αναλλακτικές λύσεις για τους αναπηρούς προκειμένου να στηρίζονται και να εξακολουθούν να ζουν μέσα στις κοινότητές τους, στους συνήθει χώρους τους. Γίνεται παραβίαση της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ανθρώπων που αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Πρόκειται για μια σύμβαση αυτή των δικαιωμάτων των αναπήρων που είναι δεσμευτική και φροντίζει ώστε να μπορούν να εξακολουθούν να ζουν στους χώρους τους, στα σπίτια του, στα άτομα με αναπηρίες. Αλλιώς καταλήγουν σε ιδρύματα και αυτό αποτελεί παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα σας δείξω πώς ζουν σε ιδρύματα ορισμένοι άνθρωποι με αναπηρίες και καταλαβαίνετε ότι οι ίδιοι είναι πιο ειδικοί για να μιλήσουν για την κατάστασή τους. Ε, δεν πρέπει λοιπόν κοινοτικά κονδύλια να πηγαίνουν σε τέτοια ιδρύματα Αντίθετα, χρειάζονται διαφορετικές δράσεις και εσείς μπορείτε να φροντίσετε γι' αυτό. Δείτε τώρα ένα πολύ σύντομο βιντεάκι. The lights. Yeah.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 da ulaže u zajednicu i da se u zajednici naprave službe podrške koje bi same osobe sa invaliditetom mogle doći i tražiti neku pomoć i uslugu koja mu u tom trenutku treba.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 čekati popune na sve svoje rupe u životu u šest godina. Znači putujem, radim, družim se, kuham. Koji sve drugi ljudi? Ceea ce văd e că statul român vorbesc de instituții ca să vadă lumea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 στο αλλά για το ναι πρέτβορη μου τι έλω πράξω ότι τρίχε ναι μα ναι κακ με κόρες με συνταγέ το να να κοινάκι λέτσι μέρε ότι έβρεψε μου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 So uh, Ζητάμε λοιπόν από την Επιτροπή σας να διατηρήσει ανοιχτή την Επιτροπή αυτή μια που έχει πάει και στην Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμών για να ελέγξει παρετέρω την κατάσταση με τα κονδύλια αυτά. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το λόγο έχει ο κύριος Ράτσμαν Μάικλ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να σχολιάσω πάνω στο θέμα αυτό. Πρόκειται για ένα ευαίσθητο και περίπλοκο ζήτημα. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει εξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα τελευταία πέντε χρόνια περίπου και είναι δύσκολο τώρα μέσα σε λίγα λεπτά να σας παρουσιάσω τα κύρια ζητήματα και τα διάφορα βήματα τα οποία έχουμε ακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο πρώτα απ' όλα και για την επόμενη μετά. Πάντως αν θέλετε ευχαρίστως να σας στείλω γραπτά περισσότερες λεπτομέρειες εξηγώντα τι ακριβώς σημαίνει αυτό στην πράξη. Πρώτα απ' όλα λοιπόν όσον αφορά την ε, πολιτική που αναπτύσσουμε στον τομέα αυτό πρόσφατα, από το 2008-2009 δεν απατώμε, αρχίσαμε με τον τότε Επίτροπο για την Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις, τον κύριο Σπίτλα, ο οποίος ετοίμασε έκθεση, ζήτησε έκθεση από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων όσον αφορά την μετάβαση από την ε, φροντίδα που δινόταν σε ιδρύματα σε φροντίδα που να δίνεται σε κοινότητες. Πρόκειται λοιπόν για μια μετάβαση που άρχισε τότε. Υπήρξε έκθεση το 2009. Στη συνέχεια βέβαια αυτό είχε κάποιες επιπτώσεις στα διορθωτικά ταμεία. Διότι στην τρέχουσα περίοδο που άρχισε το 2007 διάφορες χώρες είχαν χρήματα που τα είχαν προγραμματίσει για το κοινωνικό τομέα, τον τομέα της υγείας και η Γενική Διεύθυνση Ρέγγιο ήθελε τα χρήματα αυτά να χρησιμοποιηθούν όσο γίνεται περισσότερο για τη μετάβαση αυτή από τα ιδρύματα στην κοινότητα. Υπάρχουν ε, χώρες που αναφέρει στην αναφορά της η αναφέρουσα, η οποία βέβαια έχει δραστηριοποιηθεί ιδιαίτερα, κυρίως για τη Βουλγαρία και την Ουγγαρία, που αναφέρονται ρητά στην αναφορά, προκειμένου εκεί προγράμματα τα οποία στηρίζονται στην τρέχουσα περίοδο από τα διαστρωτικά ταμεία να αλλάξουν. Στη Βουλγαρία, για παράδειγμα, έγιναν πολλές συζητήσεις με τις εθνικές αρχές και η Βουλγαρία ε, προχωράει σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση απέναντι στα παιδιά καταρχήν, που αναφέρεται και στην αναφορά για παιδιά που βρίσκονται σε ιδρύματα, προκειμένου να κλείσουν τα ιδρύματα αυτά και να γίνει μετάβαση αυτή σε φροντίδα μέσα στην κοινότητά τους. Αυτό βέβαια μέσα σε ένα ορίζοντα 15 ετή γιατί πρέπει να ετοιμαστούν τα κατάλληλα σπίτια, οι κατάλληλες κοινωνικές υποδομές για να μπορεί να βρεθεί αυτός ο νέος τρόπος ζωής των ατόμων με αναπηρίες μέσα στις κοινότητές τους. Για την Ουγγαρία, την οποία γνωρίζει πολύ καλά η αναφέρουσα, και εκεί γνωρίζουμε ότι υπάρχουν εξελίξεις στον τομέα της μετάβασης αυτής. Η Επιτροπή έχει αναλάβει δράση ήδη από το 2009. Είδαμε ότι όντως δεν υπήρχε επαρκή στρατηγική σχετικά με την ιδρυματοποίηση στην Ουγγαρία και συστήσαμε οι Ουγγρικές αρχές να ετοιμάσουν ένα στρατηγικό πρόγραμμα ώστε να αλλάξει η κατάσταση αυτή συμμετείχαν ε, και οι υπηρεσίε μα σε σεμινάρια στην Ουγγαρία. Ζητήσαμε και την άποψη των εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι έχουν, δούλεψαν προηγουμένως στην ομάδα αυτή ad του Επιτρόπου Σπίτλα, για την οποία σας μίλησα πριν. Και συνεργαζόμαστε με τις αρχές της χώρας, προκειμένου τα κονδύλια που πηγαίνουν στην Ουγγαρία να χρησιμοποιηθούν για την αλλαγή αυτή από την ιδρυματοποίηση στις κοινότητες. Υπάρχει ένα ειδικό σώμα τώρα στη χώρα αυτή, το οποίο συμμετέχει στην εταιρική σχέση που έχουμε με την Management Authority για να συνεργαζόμαστε με την Ουγγαρία. Αυτή είναι η κατάσταση στην τρέχουσα περίοδο. Τώρα υπάρχουν και πολλές δραστηριότητες για να προωθήσουμε αντίστοιχες δράσεις και στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Η νέα ρύθμιση για τα εξωτικά ταμεία έχει ειδική διάταξη που μιλάει για χρηματοδότηση υποδομών στον τομέα της υγείας που συνεισφέρουν στην μετάβαση από την ιδρυματοποίηση στη ζωή στην κοινότητα. Ξέρω ότι πολλοί από εσά παρακολουθούν το πακέτο των δημοτικών ταμείων για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Ξέρετε ότι υπάρχει εξάντε ε, προϋπόθεση προκειμένου να εκταμιεύονται τα κονδύλια αυτά. Και υπάρχει λοιπόν τέτοια ρύθμιση που έχει να κάνει με την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. είναι κάτι που πρέπει να σέβονται τα κράτη-μέλη για να χρησιμοποιούν τα κονδύλια μας στο μέλλον. Άρα είναι ένα βήμα προς τα μπρος. Δεν υποστηρίχθηκε πλήρως το Συμβούλιο, γίνονται διαπραγματεύσεις, το Κοινοβούλιο το στηρίζει όπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οπότε ελπίζουμε ότι θα προχωρήσουμε. Χρειάζεται βέβαια νομοθετική βάση και κατευθυντήριες γραμμές για να δούμε στην πράξη πώς θα τεθούν σε εφαρμογή όλα αυτά. Και εδώ υπάρχουν δύο θέματα. Έχουμε τις κατευθυντήριες γραμμές που έχουμε ήδη ετοιμάσει όσον αφορά την φροντίδα σε κοινότητε και υπάρχει και ένα άλλο έντυπο για την χρήση των κονδυλίων από τα διαφορετικά ταμεία. Είναι πράγματα τα οποία έχουν υπογράψει οι επίτροποι και αναγνωρίζουν ότι είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει πολύ τις συζητήσεις στο μέλλον. Επιπλέον όμως ετοιμάζουμε και τις δικές μας εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές για να δούμε πώς θα τεθούν σε εφαρμογή όλα αυτά. Δεν είναι εύκολο το πράγμα, αλλά πρέπει να δούμε πιο συγκεκριμένα τι σημαίνουν οι νομικές διατάξεις της σύμβασης, αν σημαίνει ότι όλα τα ιδρύματα πρέπει να μην χρηματοδοτούνται, αν υπάρχουν ε, εξαιρέσεις, έκτακτες περιπτώσεις κλπ. κλπ. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να κοιτάξουμε πάρα πολύ σοβαρά και αυτό ακριβώς κάνουμε αυτή την περίοδο. Τέλος, για να επανέλθω στις περιπτώσεις που αναφέρονται για τη Ρουμανία και την Σλοβακία. Που αναφέρονται στην αναφορά. Ζητήσαμε από τις αρμόδιες αρχές και την Management ε, Unit να μας εξηγήσουν τι ακριβώς συμβαίνει εκεί με τα άτομα με αναπηρίες και περιμένουμε πληροφορίες ακόμα από τη Σλοβακία. Για τη Ρουμανία έχουμε 50 προγράμματα περίπου που έχουν ως ομάδα στόχο τα άτομα με αναπηρίες και είναι δύο κατηγορίες. Υπάρχουν κοινωνικά κέντρα που έχουν βέβαια πολυδιάστατες λειτουργίες και υπάρχουν και βελτιώσει που γίνονται με τη δημιουργία κοινοτικών κέντρων για τα άτομα με αναπηρίες. Εκφράζονται ανησυχίες ότι στα μεγάλα ιδρύματα γίνονται παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κακή μεταχείριση. Εμείς δεν έχουμε καμία απόδειξη ότι τα ιδρύματα τα οποία χρηματοδοτούμε προχωρούν σε τέτοιες πρακτικές. Αν υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες, η αναφέρουσα θα πρέπει είτε να πάει στην Management Authority που είναι υπεύθυνη για αυτό το θέμα και να την ενημερώσει ή αλλιώς μπορεί να στείλει προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά με συγκεκριμένα στοιχεία για προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πιστεύει ότι παραβιάζουν την, ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την νομοθεσία κλπ. Με συγκεκριμένα ονόματα ιδρυμάτων. Ευχαριστώ. Η κυρία Ντανόκα. Yes, thank you. Ευχαριστώ. Καταρχάς, να ευχαριστήσω την αναφέρουσα Νομίζω ότι αυτή η αναφορά είναι ένα πολύ σημαντικό επιχείρημα για μας ώστε να μπορέσουμε να παλέψουμε για μια οριζόντια οδηγία για μη διακριτική μεταχείριση και κυρίως για τα άτομα με αναπηρία. Δεν υπάρχει ακόμα μέχρι τώρα αυτή η οδηγία και βεβαίως το πρόβλημα δεν είναι η Κομισιόν γι' αυτό, είναι το Συμβούλιο που δεν θέλει να υπάρξει μια τέτοια οδηγία. Ε, να βερόμαστε συνέχεια στην ε, Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, αλλά δεν μπορούμε να αναφερθούμε σε κάτι δικό μας, σε μια δική μας νομοθεσία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Συμφωνώ για την αιρεσιμότητα που μπορεί να ισχύσει και για τα διορθωτικά ταμεία και συμφωνώ και με τις προσπάθειες που έχει κάνει η Κομισιόν, αλλά δεν κατάλαβα. Ε, η Κομισιόν μίλησε για την Ουγγαρία, για τη Ρουμανία. Είναι επιλεκτική η προσέγγισή σας ή ασχολείστε με όλα τα κράτη-μέλη. Έχετε επαρκή μέσα για να εφαρμοστεί αυτή η αρεσιμότητα σε όλα τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Και πρέπει να φύγω, πρέπει να πάω στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να πω και εγώ δύο πράγματα. Είμαι ε, ογκρικής καταγωγής, είμαι ψυχίατρος και πρώην υπουργό Κοινωνικών Υποθέσεων. Το σημαντικό εδώ και από ιστορικής πλευράς είναι ότι σε πολλές ε, κεντρο, ε, κεντρικές, χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και της Ανατολικής Ευρώπης ήταν σύνηθες να μπαίνουν οι άνθρωποι αυτοί σε ιδρύματα με αναπηρία είτε με ψυχολογικά προβλήματα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό για τις χώρες αυτές να επενδύσουμε τα διαρθρωτικά μας κονδύλια σε κοινοτική πρόνοια γιατί δεν υπήρχε τίποτα ανάμεσα. Είτε θα πήγαιναν σε οικογένειές τους αυτοί οι άνθρωποι χωρίς βεβαίως καμία βοήθεια από το κράτος ή θα πηγαίνανε σε κάποια τεράστια πρόσωπα ιδρύματα ανάμεσα δεν υπήρχε τίποτα. Και βεβαίω σε αυτά τα ιδρύματα υπήρχαν τεράστιε παραβιάσει θεμελιωδών δικαιωμάτων. Οι, οι εικόνε αυτέ το δείχνουν ξεκάθαρα. Δείχνουν ποιο είναι το πρόβλημα με τα ιδρύματα αυτά. Οπότε νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό η εκ των προτέρων αιρεσιμότητα και από την αρχή τα κράτη-μέλη να έχουν μια στρατηγική ε, και να μπορούν να την αποδείξουν για αυτά τα ιδρύματα πριν εγκριθούν τα, διαρθρωτικά κονδύλια που θα, τις, ε, που θα τους δοθούν για να δαπανηθούν για τέτοια θέματα. Αλλά εξίσου σημαντικό είναι και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. Αν ρωτήσει κανείς ε, στις χώρες αυτές τους πολίτες, οι περισσότεροι θα σας πούν ότι αυτή είναι η λύση, να επενδύσει κανείς σε αυτά τα τεράστια ιδρύματα. Θυμάμαι όταν έκανα εγώ κάποιες ε, συναντήσεις με διάφορους δημάρχους που τους ε, ζητούσαν να μου πούνε το όραμά τους, το όνειρό τους για, για το πώς θα χρησιμοποιήσουν τα ε, κονδύλια. Και όλοι έλεγαν ότι θα ήταν τέλειο αν μπορούσαμε να έχουμε ένα μεγάλο ίδρυμα που θα φροντίζει ανθρώπους με ψυχολογικά προβλήματα ή με αναπηρίες, γιατί έτσι μπορούσαν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας για την κοινότητά τους. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με αυτό και είναι σημαντικό να υπάρξει διαφάνεια ω προς αυτό, να υπάρχουν δηλαδή συγκεκριμένα δεδομένα πραγματικά για το τι γίνεται και πώς δαπάνονται τα κονδύλια, αν η δαπάνη τους είναι σύμφωνη με την σύμβαση των, του ΟΗΕ, με την οδηγία για τη μη διακριτική μεταχείριση κτλ. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ θεμητό, μια πολύ θεμητή πρωτοβουλία να το παρακολουθήσουμε, να παρακολουθήσουμε τι ακριβώς γίνεται σε αυτές τις χώρες σε ό,τι αφορά τη δαπάνη των διαρθρωτικών κονδυλίων. Οπότε ζητώ από την Κομισιόν να μα δώσει τα δεδομένα και να είναι πολύ αυστηρή σε ό,τι αφορά την ε, εκ των προτέρων ε, ρεσιμότητα, να παρακολουθήσει πολύ στενά την δαπάνη αυτών των ε, κονδυλίων και να δώσει βεβαίω την βοήθεια που χρειάζεται. Δεν μπορούμε να επαφιέμεθα πάντα στην καλή θέληση των κρατών μέσω αυτής της κινητοποίησης ε, ε, των, τοπικών τοπικών κοινωνιών. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη ως προς αυτό. Σας ευχαριστώ και βεβαίως θα το υποστηρίξω να έχουμε δεδομένα και ελπίζω να μπορέσει αυτό να περάσει και για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό ταμείο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να τονίσω διάφορα θέματα. Η συνάδελφος είπε ότι δεν ε, έχουμε δική μας ε, ρύθμιση. Ναι, με τις Ηνωμένα Έθνη έχουμε υπογράψη και έχουμε ένα το νομικό μέσο, αλλά η Σύμβαση των Μεδεθνών αποτελεί μια αναφορά και εκεί στο μέλλον θα πρέπει να βασιστούμε. Η σχετική προϋπόθεση ήταν ε, αυτό περί μη διάκρισης. Ε, τι σημαίνει αυτό είναι οι νέε δημοσιονομικέ προοπτικέ. Εκεί μέσα βρίσκεται και τα καλά ριζωμένο και ε, ίσως όμως χαθούν και κονδύλια εάν δεν βασιστούν στη συνθήκη και διαφορετικά όμως αν δεν μπορούμε να προσαρμοστούμε δεν θα μπορούσαμε να βασιστούμε και στη Σύμβαση των Εθνών. Όταν είδα αυτή την ε, βίντεο, αυτό το βίντεο ε, προσπάθησα να καταλάβω γιατί πέρα από κάθε δράση υπάρχουν άτομα και είδαμε την ε, ε, Ρουμένα, την Κροάτισσα και βλέπουμε ότι διάφορα πραγματικά συμβαίνουν εδώ. Το θέμα παραμένει, να παραμείνει εκρεμές, ανοιχτό και να δούμε ε, ότι ακριβώς δεν είναι σωστό αλλά συμβαίνει και θα πρέπει να δούμε πώς θα υποστηρίξουμε τα βασικά δικαιώματα και να μην ε, ε, είμαστε υπέρ αυτής της παρεμβίωσης των δικαιωμάτων ατόπων με αναπηρίες και πολλοί ζητούν μια ανεξάρτητη ζωή και το βλέπουμε και με άλλους αναφέροντες ε, όπως και οποιοδήποτε, οποιοδήποτε άλλη ανθρώπινη ύπαρξη όταν έχει τις δραστηριότητες του σε διάφορους δεκάδες τομείς να μπορεί να οργανώσει τη ζωή του με πλήρη ανεξαρτησία, αλλά έχουμε και διάφορες βαριές αναπηρίες που σημαίνει ότι θέλουν κατοίκον φροντίδα. Και όλο αυτό αποτελεί μια διαδικασία, γιατί εντάξει μια ελαφρά αναπηρία με κάποια βοήθεια φτάνει, αλλά μια βαριά αναπηρία θα χρειαστεί και ένα καταλληλό κέντρο και μια εξειδίκευση και ίσως να παραμείνει εγκλειστός κάπου. Και σε μερικές φορές ε, θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε όμως μια μια ανεξάρτητη ζωή. Όλα αυτά έχουν να κάνουν και με οικονομικά θέματα για να καταστεί δυνατό. Και καταλαβαίνουμε το πόσο ανησυχούν ε, και τα μέλη λόγω και της οικονομικής κρίσης, λόγω της ύφεση στην Ευρώπη. Εκεί δυστυχώς να, πρέπει να προσέξουμε να μην θυγεί καμία πρόοδος που έχει ήδη επιτευχθεί γιατί βλέπουμε ότι περικόπτεται συντάξεις ε, και βλέπουμε ε, να μην, δεν πρέπει να κλείσουν κέντρα υποδοχής αναφύρων. Δεν θα πρέπει να θίξει το δικαίωμα προσεργασία αυτών των ατόμων με αναπηρία, γιατί τότε θα έχουμε χάσει πολλά καθοδόν και θεωρώ ότι σε παρόμοιες στιγμές κρίσης εκεί είναι που θα πρέπει να προσταθούν οι ίσες ευκαιρίες, ίσες ευκαιρίες για όλους και ακριβώς θα πρέπει πραγματικά να κάνουμε αυτά που πιστεύουμε, αυτά που υποσυπογράψαμε και στα Ηνωμένα Έθνη και με με τη σύμβαση ακριβώ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μπάγκο, κύριο Μπάγκο. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα ξεκινήσω λέγοντας, όπως και η κυρία Γκένς, να σας πω, είμαι ούγκρο, είμαι νομικός και διεύθυνα ε, σε ένα, ένα δήμο ε, παρόμοια κέντρα και αν ρίξουμε μάτια στο βαθμό ανάπτυξης και κοινωνικής ευαισθησίας μιας χώρας, όλα αυτά πραγματικά περιγράφονται, δείχνονται μάλλον με τον τρόπο που ασχολούνται και αντιμετωπίζουν τους ανάπηρους και τις, τα διάφορα κέντρα. Και ο κύριος Κούσα όπως ζήτησε, ζήτησε πληροφορίες για ανάπηρο που είναι πολύ σημαντικό στην αναφορά αυτή να δούμε ότι για την Ουγγαρία και τη Βουλγαρία διαφέρει κάπως η κατάσταση από τη μεταξύ Ρουμανίας και Βουλγαρίας και Επιτροπή είπε ότι έχουν παρουσιαστεί νέα στοιχεία από το 2009 από το Δασπίντλα που ε, ήδη κάτι καινούριο συστάθηκε και μια νέα στρατηγική για 30 ολόκληρα χρόνια για τον κόσμο που υποφέρει από παρόμοιες αναπηρίες. Και με τον νέο νόμο τι προβλέπετε, ότι δεν μπορούν τα κέντρα να υποδεχτούν πάνω από 50 άτομα και τα κέντρα αυτά πραγματικά στην Ουγγαρία δεν έχουν πάνω από 50 άτομα. Και για τις μεταβολές ε, για αυτά τα κέντρα σε 15-20 κέντρα έχουμε 1500 περίπου άτομα και θα βελτιωθούν οι συνθήκες υποδοχής τους τα προσεχή χρόνια. Κάπως λοιπόν άλλαξε η κατάσταση και αυτό η αναφορά ήταν το 2008-2009 και τότε η Ουγγρική κυβέρνηση ήθελε, εξ, μάλλον, ε, ανεκκίνωσε την άποψή της και τη θέση της ότι θα ξόδευε αρκετά εκατομμύρια φιωρίνια τοπικό νόμισμα για τα κέντρα αυτά. Και εδώ μεταξύ, επαναλαμβάνομαι, αυτά ξεκίνησαν το 2009 με αυτή την αναφορά και για τη Βουλγαρία και την Ουγγαρία τώρα δεν ισχύει πια αυτή η αναφορά. Για τη Σλοβακία δε εξετάζει το πως έχει κατάσταση η Επιτροπή και στη Ρωμανία λόγω της θέσης του Συμβουλίου και της ίδιας ε, της ρουμανικής κυβέρνησης η άποψή μας ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε πάντως να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά αυτή και από νομικής πλευράς θεωρώ ότι για τη Ρουμανία πρόκειται για θέμα, για πρόβλημα σημαντικό. Θα πρέπει επαναλαμβάνω να παραμείνει ανοιχτό το θέμα αλλά διαδικαστικά περιλαμβάνει και άλλα κράτη. Δυστυχώς ε, δεν ξέρω κατά πόσο εξουδετούμεθα να συνεχίσουμε την εξέταση. Θα πρέπει να κλείσει όμως αυτό εδώ και να επανέλθουν οι αναφέροντες με μια νέα πρόταση, με μια νέα αναφορά που να αφορά τη Ρουμανία. Ο κύριος Μαρτίνας Μαρτίν. Ευχαριστώ. Αυτό είναι ένα θέμα ιδιαίτερα περίπλοκο. Νομίζω ότι όλοι συγκινούμαστε, μας δημιουργεί αίσθηση ένα βίντεο σαν και αυτό που είδαμε πριν από λίγο. Εξάλλου είναι ένα θέμα που τουλάχιστον πολλούς από εμά μας αγγίζει και προσωπικά. Και αυτό γιατί γνωρίζουμε ανθρώπους. Εγώ προσωπικά γνωρίζω αρκετούς ανθρώπους που η καθημερινή τους ζωή επηρεάζεται από αυτή την κατάσταση. Εμένα συγκεκριμένα προσωπικά. Και όλοι έχουμε στον περίγυρό μας, πιο κοντά ή λιγότερο κοντά, κάποια άτομα με αναπηρίες. Και σκέφτομαι το εξής. Οι πληροφορίες που μας έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σίγουρα είναι ενδιαφέρουσες και με καθησυχάζουν κάπως, στο βαθμό δηλαδή που Καταλαβαίνω ότι είναι στην ημερήσια διάταξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν αγνοεί δηλαδή το ζήτημα αυτό η Επιτροπή. Ωραία. Διαπιστώνω όμως ότι, όπως συμβαίνει και με άλλα πράγματα, και εδώ η κατάσταση διαφέρει από χώρα σε χώρα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως ακριβώς γιατί προερχόμαστε από διαφορετικά συστήματα. Άρα η προσέγγιση που θα ακολουθήσουμε μπορεί να είναι κάπως διαφορετική αν και βασίζεται σε πολύ συγκεκριμένες αρχές. Αυτό που έχει σημασία είναι να εξυπηρετεθούν όλες οι περιπτώσεις και να είμαστε συγχρόνως ρεαλιστές στο πώς θα εφαρμόσουμε αυτές τις αρχές που αποφασίζουμε. Στη χώρα μου, αλλά και σε άλλες χώρες του περιγυρού μου που γνωρίζω καλά, προερχόμαστε από μια κατάσταση όπου τα 30 τελευταία χρόνια εντοπίστηκαν δικαιώματα για ομάδες που προηγουμένως δεν είχαν τα δικαιώματα αυτά. Πριν από 40 χρόνια δηλαδή τα άτομα με αναπηρίες δεν είχαν κανένα δικαιώμα. Τους παρκάραμε βασικά κάπου. Ποτέ δεν είχαμε φανταστεί τότε ότι η κατηγορία αυτή ατόμων θα μπορούσε να έχει δικαιώματα, ιδιαίτερα δικαιώματα ενώ πρόκειται για πολίτες βέβαια. Ξαφνικά εμφανίστηκαν λοιπόν τα δικαιώματα αυτά, όπως και τα δικαιώματα της γυναίκας που δεν υπήρχαν τότε ή τα δικαιώματα των ομοφιλόφιλων και πολλών άλλων ομάδων που υπέφεραν από διακρίσεις σε βάρος τους από την κοινωνία για αιώνες. Σιγά σιγά λοιπόν η κοινωνική πρόοδος στην Ήπειρό μας βοήθησε ώστε να εντοπιστούν και να εμφανιστούν δικαιώματα ομάδων που νωρίτερα δεν αντιμετωπίζονταν επίσης όρις με τους υπόλοιπους πολίτες. Και αυτό μέσα βέβαια από συνταγματικά κείμενα, αλλαγές ε, στη διεθνή κοινότητα κτλ. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε με τα δικαιώματα αυτά και να τα κάνουμε ακόμα πιο συγκεκριμένα. Σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός εξαίρεσης, πρέπει να ξέρουμε ότι ήταν οι ίδιοι, τα ίδια τα θύματα κατά κάποιο τρόπο, οι οποίοι φρόντισαν να αναγνωριστούν τα δικαιώματά τους. Οι γυναίκες, για παράδειγμα, ήταν εκείνες οι οποίες φρόντισαν να αναγνωριστούν τα δικαιώματά τους. Οι ομοφιλόφιλοι ήταν εκείνοι οι οποίοι φρόντισαν να αναγνωριστούν τα δικά τους συλλογικά δικαιώματα. Και τα άτομα με αναπηρίες τα ίδια φρόντισαν να αναγνωριστούν τα δικά τους τα δικαιώματα και να το μάθουμε και εμείς αυτό, επειδή ακριβώς έχουμε κάποιους στον περίγυρό μας. Υπάρχει όμως κάτι το οποίο με ανησυχεί ιδιαίτερα στην αναφορά που εξετάζουμε σήμερα. Εννοείται ότι συμφωνώ και εγώ να παραμείνει ανοιχτή και να συνεχίσουμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτήν. Είναι ένα θέμα που χρειάζεται την δικιά μας βοήθεια και προσπάθεια. Αλλά υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Το θέμα δεν είναι να καταργήσουμε μηχανισμούς, αλλά να φροντίσουμε οι μηχανισμοί αυτοί να είναι συμβατοί. Το είπε και κάποιο που μίλησε πριν από μένα. Είναι προφανώς, είναι προφανές, συγγνώμη, ότι η αναπηρία έχει διαφορετικές διαβαθμίσεις. Υπάρχουν αναπηρίες που δεν έχουν άλλες λύσεις πέρα από τα ιδρύματα αυτά, τα κέντρα αυτά. Βέβαια εννοείται ότι τα κέντρα αυτά πρέπει να λειτουργούν με καλό τρόπο και όχι να κακομεταχειρίζονται ε, τα, τους τροφίμους τους, εννοείται. Αλλά πέρα από το θέμα αυτό του σεβασμού της αξιοπρέπειας των ατόμων με αναπηρία, τα κέντρα αυτά μπορούν να παραμείνουν σε ορισμένες περιπτώσεις. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα, το θέμα του πώς λειτουργούν αυτά τα ιδρύματα. Εννοείται ότι η κοινωνία έχει υποχρέωση να τα ελέγχει και να φροντίζει να μην παραβιάζεται ποτέ η αξιοπρέπεια των ατόμων. Δεν πρέπει να είναι κάτι σαν παρκάρισμα πολιτών επειδή έχουν αναπηρίες και είναι πολύ ευάλωτοι και δεν μπορούν να αντιδράσουν ή να υποστηρίξουν τα δικαιώματά τους. Με αυτό συμφωνούμε νομίζω όλοι. Αλλά το πραγματικό πρόβλημα είναι, μάλλον το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι να πούμε όχι, όχι, οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχουν άλλοι τρόποι φροντίδας και να καταργήσουμε τα ιδρύματα. Όχι, και τα ιδρύματα μερικές φορές είναι αναγκαία. Και η μία δομή και η άλλη. Όπως στη χώρα μου για παράδειγμα, καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι αναγκαίο ο νόμος της ε, εξάρτησης που τι έλεγε. Έλεγε ότι πρέπει να παίρνουν κάποια χρήματα. Το 90% ήταν οι γυναίκες ε, στις οικογένειες που φρόντιζαν κάποιο άτομο με αναπηρία, γιατί μέχρι τότε το κάνανε εντελώ δωρεάν. Όμως όχι, τα άτομα τα οποία φροντίζουν για κάποιον με σοβαρή αναπηρία πρέπει να αναγνωρίζεται από τις κρατικές αρχές και να μείβεται γι' αυτό. Στη χώρα μου, λοιπόν, υπάρχουν δημόσια ιδρύματα, υπάρχουν όμως και ιδιωτικά. Υπάρχουν δηλαδή μονάδες κοινωνικού χαρακτήρα που μπορεί να έχουν θρησκευτική προέλευση ή συνεταιριστικά ιδρύματα που έχουν φτιάξει ίδιες οικογένειες ή τα ίδια τα άτομα με αναπηρίες. Και κάποια από αυτά τα κέντρα λειτουργούν πολύ ικανοποιητικά. Και άλλα τα οποία δεν λειτουργούν ικανοποιητικά. Αυτό λοιπόν το οποίο με απασχολεί εδώ και με ανησυχεί κάπως είναι αυτό που λέει η αναφορά, ότι δηλαδή πρέπει να είναι παράνομο το να χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση κάποιο από αυτά τα τρία διαφορετικά είδη φροντίδας. Είπαμε, είναι είτε η οικογενειακή βοήθεια, είτε τα ιδρύματα, είτε η βοήθεια τα κονδύλια, δηλαδή για να ζουν οι ανάπηροι μέσα στις κοινότητές τους. Υπάρχουν τρεις διαφορετικές δυνατότητες. Δεν πρέπει να πούμε ότι είναι παράνομη χρηματοδότηση καμιάς από τις τρεις αυτές κατηγορίες φροντίδας. Πρέπει να είναι συμβατές μεταξύ τους, να μπορούν να συνεπάρχουν. Γιατί και στις τρεις περιπτώσεις μπορεί να εντοπίζει κανείς ε, κακή λειτουργία, δεν λέω. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν, δεν πρέπει να τις αγνοούμε, πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε επίσης ότι και στις τρεις περιπτώσεις υπάρχουν και αξιόλογες προσπάθειες και αξιοπρόσεχτη λειτουργία που πρέπει να σεβαστούμε και να στηρίξουμε. Γι' αυτό λοιπόν η αναφορά που εξετάζουμε σήμερα που είναι για ένα πολύ σοβαρό θέμα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή και να εξακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ενημερώνει για την πρόοδο που έχουμε στην εξέταση του ζητήματος αυτού. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριο Πάσκα. Euh, Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το πώς λειτουργούν οι κοινωνικές υπηρεσίες για τα ανάπηρα άτομα σε Ρουμανία, Βουλγαρία και Ουγγαρία δεν το γνωρίζω, δεν τη γνωρίζω αυτή τη λειτουργία. Αλλά η Επιτροπή έκανε μια εκτίμηση αυτών των παροχών στη Σλοβακία και είπε ότι πρόκειται για ένα καλό παράδειγμα σωστής ενέργειας Βέβαια θα μπορούσαμε ακόμα περισσότερο να κάνουμε στη χώρα μου για τους ανάπηρους, για τα άτομα με αναπηρία. Η σλοβακική κυβέρνηση είμαι σίγουρος ότι θα χρησιμοποιήσει κάθε δυνατό μέσο για να βελτιώσει αυτές τις υπηρεσίες για άτομα με αναπηρίες. Αυτά και σας ευχαριστώ. Äh, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους αναφέροντες. Συμφωνούμε νομίζω ότι το θέμα αυτό πραγματικά είναι πολύ σημαντικό και μάλιστα πολλά από ήθελα να πω τα είπαν οι προλαλήσαντες. Αν θέλουμε όντως να κινητοποιήσουμε την, την κοινωνία, αν θέλουμε να αλλάξουμε στην κοινωνία το πώς αντιμετωπίζει η ίδια η κοινωνία το, τα, τα άτομα με αναπηρία, πρέπει όντως να δράσουμε. Θέλουμε να τους ενσωματώσουμε στην, ε, στην κοινωνία. Και στη δική μου την χώρα τώρα γίνονται πολλές προσπάθειες αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να πηγαίνουν στα σχολεία που πηγαίνουν και όλοι οι υπόλοιποι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είναι πραγματικά, ε, θα, θα μπορούν έτσι να είναι κομμάτι της κοινωνίας. Γι' αυτό πρέπει να πω ότι είμαι ε, υπέρ του να παραμείνει ανοιχτή η ε, αναφορά αυτή έτσι ώστε να μπορούμε να την παρακολουθήσουμε. Γιατί πάντα η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Ε, και υπάρχουν και κάποιες δυνατότητες που έχουμε για το πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε τους ανθρώπους αυτούς. Ε, το πρώτο είναι η οικογένεια. Όταν λειτουργεί η οικογένεια μπορεί να ε, εγγυηθούμε την ενσωμάτωσή τους και στην ευρύτερη κοινωνία. Μετά μπορούμε να τους δώσουμε δική τους, ε, δικό τους, ένα δικό τους σπίτι έτσι ώστε να μπορούν να έχουν και αυτή τη δική τους ύπαρξη, να μην εξαρτώνται πάντα από κάποιον. Βεβαίω θα μπορούμε να τους δώσουμε και μια βοήθεια. Μπορεί κάποιο να είναι εξάρτητο, αλλά να μπορεί να στηριχτεί και σε κάποιον. Ε, δεν είναι ίδρυμα αυτό, αλλά θα μπορούσαμε ε, να, να προσφέρουμε μια βοήθεια στους ανθρώπου αυτούς. Και κάτι άλλο είναι όντως ε, αυτή η η εγκατάστασή του σε ε, ιδρύματα. Βεβαίω, αυτό θα εξαρτηθεί και από την περίπτωση του κάθε ανθρώπου. Σημαντικό όμως είναι να προσέχουμε πάντα οι άνθρωποι αυτοί με αναπηρίες ε, να έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν μέρος στην κανονική ζωή της κοινότητας, έτσι όπως έχουμε και εμείς την ε, δυνατότητα να παίρνουμε μέρος στη ζωή της κοινότητάς μας. Είναι σημαντικό λοιπόν να το παρακολουθήσουμε, θα ήταν λάθος μήνυμα να, το, να κλείσουμε την αναφορά αυτή, ε, ακριβώς για σκοπούς παρακολούθησης. δεν είναι το θέμα μόνο των χωρών που αναφέρονται στην αναφορά. Το θέμα της πνευματικής αλλαγής των ανθρώπων είναι θέμα όλης της Ευρώπης. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να παραμείνει ανοιχτή αυτή η ε, αναφορά. Είναι πάρα πολύ λογικό, είναι σκόπιμο για να... και βεβαίω θα μπορούσαμε να τη δώσουμε και στις καθόλου αρμόδιες επιτροπές να τη μελετήσουν γιατί είναι θέμα πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι ε, πρέπει να παρακολουθήσουμε το τι θα γίνει από εδώ και μπρος και αν υπάρξουν έτσι κάποιες, ε, κάποια προβλήματα στην όλη διαδικασία να μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε για να τα λύσουμε. Ο κύριος Μπάγκο. Ε, ε, ναι, κυρία Πρόεδρε, με τους συναδέλφους συνοηθήκαμε, συζητήσαμε Εάν αυτός ο έλεγχος μπορεί να ασκηθεί σε όλες τις χώρες, τότε επανερχόμαστε στο δική μου άποψη και θα θέλαμε να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά και να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε και με την νομική υπηρεσία της Επιτροπής και να παρακολουθήσουμε θα αλλάξει τη θέση του το Συμβούλιο ναι ή όχι. Τότε μπορούμε να συμφωνήσουμε και να έχουμε μια κοινή δράση. Ναι, ένα λεπτό ο αναφερόμενος για να... ο αναφέρον για να μας δώσει την απάντηση, για να μας δώσει την απάντησή της. Ευχαριστώ πολύ για όλα αυτά τα σχόλιά σας που στηρίζετε την αναφορά μου. Ακούω ότι έρχεται η αναφορά αυτή από τα άτομα που βρίσκονται σε ιδρύματα. Ε, πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να δείξουμε ότι δεν είναι έτσι. Δεν πρέπει έτσι καλλιώς να υπάρχει διάκριση. Τα άτομα με αναπηρίες δεν πρέπει να βρίσκονται μέσα σε ιδρύματα και ο βαθμός ε, αναπηρίας τους είναι άσχετος. Πρόκειται για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κανένας από μας δεν θέλει να νιώθει υποχρεωμένος να ζει χωριστά από την υπόλοιπη κοινωνία ή να ζει όχι με αυτούς που θέλει αλλά να υποχρεώνεται να ζήσει με κάποιους που έχουν την ίδια αναπηρία για παράδειγμα με αυτό. Το θέμα του κατά πόσο είναι υποχρεωτικό κάποιες αναπηρίες να αντιμετωπίζονται μόνο ιδρυματικά δεν είναι αλήθεια. Εξαρτάται πάντα από το βαθμό στήριξης που θα δώσει η κοινωνία στα άτομα αυτά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ε, να βλέπουμε ότι εκφράζονται διάφορες ανησυχίες και χρειάζεται να τις προσέξουμε. Βέβαια όλοι ζητούν να παραμείνει ανοιχτή αναφορά. Αυτό και θα πρέπει να γίνει. Για μας θεωρώ ότι χρειάζεται πρώτα απ' όλα να απευθυνθούμε στις εθνικές αρχές που εμφανίζονται εδώ και στην αναφορά ότι είναι αρμόδιες και να του ζητήσουμε μία απάντηση για τις καταγγελίες οποίες προβαίνει η αναφορά για τα συστήματα, για την εθνική νομοθεσία, την εθνική ρύθμιση για το πώς φροντίζονται αυτά τα άτομα με αναπηρίες. Και αν η ακριβώς η αντιμεσόπιση τους είναι αντίθετη με τις αρχές ίσης αντιμετώπισης και ίσων ευκαιριών προς όλους τους πολίτες όπως το επιβεβαιώνουν άλλωστε και οι διάφορες συνθήκες και ο χαρτής θεμελιωδών δικαιωμάτων και σχετικά με την χρήση ή κατάχρηση των διαχωτικών κονδυλίων στην ε, Κοκομπούνα την Επιτροπή μας να απευθύνουμε ένα ερώτημα σχετικά με την ε, χρήση των κονδυλίων σε αυτές τις ειδικέ περιπτώσεις που καταγγέλλονται και επίσης ε, στην Περιφερειακή Επιτροπή μια επαφή μαζί τους γιατί ασχολείται με τη νέα οργάνωση για τα διευθυντικά ταμεία και να τους παροτρύνουμε να προσέξουν περισσότερο τα συστήματα ελέγχου, τη διαφανή χρήση των διαφορετικών κονδυλίων όπως το είπε και ο εκπρόσωπος της Επιτροπής εδώ. Άρα λοιπόν εμείς να βοηθήσουμε με την Επιτροπή μας όλα αυτά που ακούσαμε εδώ τώρα. Και όπως το είπε και η συνάδελφος Ζανόγκα, Στη συνέχεια θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε και με την παλιότερη εργασία για την ε, οδηγία κατά των διακρίσεων, να δούμε σε ποιο σημείο βρίσκονται τα πράγματα και στην αρμόδια επιτροπή να επανεξεταστούν τα θέματα τα οποία εμείς ε, λέμε συνέχεια ότι θα πρέπει να προσεχτούν. Ευχαριστώ τους αναφέροντες, ευχαριστούμε την Επιτροπή και κλείνουμε το σημείο αυτό στην ημερήσια διάταξη. Θα πάμε τώρα, μισό λεπτό, μισό λεπτό, να ξανακάνω την πρότασή μου. Είναι όλα σωστά έτσι όπως το είπατε. Αλλά δεν θέλω να περιοριστούμε μόνο στις χώρες που αναφέρονται στην ε, αναφορά. Θέλω να, τη διευρύνουμε, να το διευρύνουμε το αίτημα, να κάνουμε μια ευρωπαϊκή συζήτηση. Βεβαίως ε, θα μπορούσαμε να βασιστούμε σε αυτά που λένε οι χώρες, οι συγκεκριμένες, ε, που είναι στην αναφορά, αλλά θέλω να, να διευρυνθεί η συζήτηση αυτή και στα 27 κράτη-μέλη. Εμείς ως Επιτροπή θα πρέπει να το ζητήσουμε να χρησιμοποιήσουμε το δικαίωμα που έχουμε. Α, συγγνώμη, συγγνώμη, 28. Εντάξει, 28, 28. Δεκτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να ε, διαβρύνουμε τη συζήτηση σε όλου, να μην περιοριστούμε μόνο στι χώρε τη αναφορά. Από τη στιγμή που συμφωνείτε, θα ζητήσουμε να γίνει έρευνα σε όλε τι χώρε τη Ένωση. Σα ευχαριστώ. Έχουμε το σημείο 9 τώρα της σημερινής διάταξης, είναι η 279 του 2012 από Ούγγρο πολίτη σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συνταξιδοτικού συστήματος που ισχύει για τα άτομα με αναπηρία στην Ουγγαρία. Ο αναφέρον δεν παρίσταται. Ο εκπρόσωπος όμως της, επι... Ε, εκπρόσωπος της Επιτροπής έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία είναι πολύ περιορισμένη. Η μόνη οδηγία που υπάρχει είναι η 2078 που απαγορεύει τη διακριτική μεταχείριση επί τη βάση διαφόρων ε, ε, κριτηρίων συμπεριλαμβανομένης και της αναπηρίας. Παρ' όλα αυτά η οδηγία αυτή εφαρμόζεται μόνο στον τομέα της απασχόληση. είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών να οργανώσουν ε, τα προγράμματα κοινωνική ασφαλισή του και η νομοθεσία του κάθε κράτου μέλου είναι αυτή που θα ορίσει τι συνθήκε σύμφωνα με τι οποίε τα επιδόματα κοινωνική πρόνοια θα δίνονται και ε, ποιο είναι το ύψο των επιδομάτων αυτών και η περίοδο για την οποία θα δίνονται συν της, ε, συμπεριλαμβανομένων και των ε, συντάξεων αναπηρία. Συμπερασματικά, η Κομισιόν λυπάται που η κατάσταση στην Ουγγαρία είναι έτσι όπω την περιγράφει ο αναφέρον, αλλά λόγω του ότι δεν υπάρχει αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά επιδόματα, κυρίω σε ό,τι αφορά το ποσό των συντάξεων, του ύψους των συντάξεων αναπηρίας, η Κομισιόν δεν μπορεί να σχολιάσει περαιτέρω αυτή την αναφορά. Η κυρία Γκιόντς. Λοιπόν, ναι, θα μιλήσω ουγγρικά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έχει να κάνει με εθνική αρμοδιότητα σχετικά με το συνταξιδοτό σύστημα. Για το... Όλα αυτά είναι βάσιμα γιατί ο τρόπος ε, που άλλαξε η κατάσταση στην Ουγγαρία για τα άτομα με αναπηρία Τη 20 Δεκεμβρίου το Κοινοβούλιο το Εθνικό υιοθέτησε, θέσπισε νόμο για τη μεταρρύθμιση του συνδεξιδοτικού συστήματος και των κοινωνικών παροχών. Και μετά αυτό τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου της επόμενης χρονιάς. Δέκα μέρες είχαν μόνο για να προετοιμαστούν αυτοί που ήταν από 57 ετών και κάτω ε, αντιμετώπισαν νέα προβλήματα ενώ εκείνοι που ήταν έτοιμοι να εξοδηθούν όχι και θα ζητούσαν κανονικά διάφορες εγγυήσεις αλλά αυτές οι εγγυήσεις ε, δεν ίσχυαν δεν υπήρχαν οι κατάλληλες εγγυήσεις στα πλαίσια του κοινωνικού ουγγρικού συστήματος και μειώθηκαν και οι συντάξεις γιατί θεσπίστηκε ένας φόρος και από τη στιγμή που που θα ισχύσει κι άλλος φόρος, τότε θα μειωθούν ακόμα περισσότερες οι συντάξεις. Και επίσης, θίγεται το δικαίωμα συνεισφόρας Ναι, χρειάζεται όλα αυτά να τα δούμε. Ε, υπάρχει και ένας έλεγχος που ασκείται και αν κάποιος δεν εμφανίζεται σε αυτόν τον έλεγχο, δεν εμφανίζεται σε αυτόν τον έλεγχο, τότε διακόπτεται η συνταξιοδότησή του. Ναι, και δεν υπάρχει και δυνατότητα προσφυγής στη συνέχεια. Και εγγράφως ε, ειδοποιούνται οι ενδιαφερόμενοι δεν υπήρξε όμως κάποια απόφαση συγκεκριμένη και να ασκήσουμε προσφυγή μας εμείς. Απλά και μόνο έλαβαν τη σχετική ανακοίνωση, τα πράγματα αλλάζουν και τίποτα άλλο. Και επίσης ε, διάφορες άλλες, διάφορα άλλα επιδόματα διεκόπησαν όπως ε, μια βοήθεια για διάφορα ταξίδια και δυνατότητες εξέβρεση εργασίας άλλης και να που ένα εμπόδιο τώρα πια και θίγονται τα κεκτημένα χάρη στην εργασία και από νομικής πλευράς αυτό που θα πρέπει να ισχύει είναι έτσι ξαφνικά προσδόκητα από μια στιγμή στην άλλη να διακόπτονται παρόμοιες παροχές τη στιγμή που ίσχυαν επί μακρό χρονικό διάστημα. Και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που ασχολήθηκα με το θέμα της υποχρετικής συνταξιοδότησης δικαστών ε, έτσι αντιμετώπισαν και αυτά τα πράγματα και Αυτό επειδή είχε αλλάξει η ηλικία ε, υποχρεωτικής ταξιδότησης, γιατί από 70 ετών υποχρεώνται τώρα να συνταξιδοθούν μόνο στα 72 αλλά και η απόφαση βασίστηκε στο ότι δεν συντάχθηκε κατάλληλα σχετική πρόταση και δεν υπήρξε δυνατότητα αντίδρασης, προσφυγής κλπ. Το ίδιο και για τα άτομα με αναπηρία. Επαναλαμβάνω, ή δεν ισχύουν πια τα επιδόματα ή τα επιδόματα μειώθηκαν κατά πολύ. Δεν υπάρχει δυνατότητα αντίδρασης, προσφυγής, γιατί όλα αυτά δεν βασίζονται σε μια συγκεκριμένη ανακοίνωση απόφασης, αλλά σε ανακοίνωση. Και βέβαια Κανονικά ένα κράτος μπορεί να καθορίζει το πώς, αλλά εδώ σημειώνεται, παρουσιάζεται πρόβλημα. Πρόβλημα και με τις συντάξεις, αλλά και με το κράτος δικαίου και με μια κάποια εγγύηση και εξασφάλιση νομική. Είναι απόντες οι αναφέροντες και γι' αυτό ακριβώς εγώ έκανα την... σας έδωσα μια περίληψη γιατί οι ίδιοι δεν μπόρεσαν να παραστούν. Μαρτίνες Μαρτίνες. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε σε αυτά που είπα προηγουμένως ε, για την προηγούμενη αναφορά βλέπω ότι ξεπερνιέται γιατί από τις μεγαλύτερες, περισσότερες προσπάθειες τις πιο θεαματικές ε, στη χώρα μου την Ισπανία πριν από 4-5 χρόνια αυτό ακριβώς για την εξάρτηση να δούμε ορισμένους μηχανισμούς, ορισμένες μεθόδους, αλλά δεν ήταν μπορώ να πούμε συντάξεις ήταν μια κάποια αμοιβή, ένα κάποιο επίδομα ώστε οι εργαζόμενοι να μπορέσουμε να τους ανταμείψουν όπως πρέπει και αξιοπρεπώς ακριβώς. Η προσπάθεια αυτή ο νόμος αυτός που αποτέλεσε και πυλώνα των προσπαθειών της κυβέρνησης στην Ισπανία μερικές φορές ε, δεν είχε τα απαραίτητα κονδύλια ας πούμε. Άρα λοιπόν ήταν μεν σημαντική ε, χειρονομία αλλά χρειαζόταν ε, παραπάνω προσοχή. Εδώ ακριβώς είπε ο προηγούμενος ομιλητής ότι η κρίση δεν θα έπρεπε πουδενή να θίγει την όλη πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις χώρες μας σχετικά με θέματα προστασίας παρομοίων ομάδων που αντιμετώπιζαν παραδοσιακά διακρίσεις και προβλήματα όπως είναι ακριβώς η κοινωνική ομάδα των ατόμων με αναπηρία και εκείνων ε, που δεν είναι εξαρτώμενοι αλλά τουλάχιστον ε, έχουν την ευθύνη να σφροντίζουν. Νομίζω ότι το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Να υποβάλω μία πρόταση. Η αναφορά να παραμείνει ανοιχτή αλλά η Επιτροπή να μπορέσει να προσπαθήσει να συνταχθεί μια λεπτομερής έκθεση, μελέτη για να δούμε πώς ακριβώς, με ποιο τρόπο επηρεάζει τα πράγματα η κρίση, τις υπηρεσίες, τις συντάξεις, όλες αυτές τις προσπάθειες που καταβάλαμε αυτά τα χρόνια στις κοινωνίες μας και ταυτόχρονα να δούμε το πρότυπο το κοινωνικό, την εξέλιξη την κοινωνική

βλέπουμε ότι χάνουν έδαφος ε, ενώ κανονικά προσπαθούσαμε να βοηθήσουμε άτομα με αναποηρία είτε τους όσους ασχολούνται με αυτούς ε, να τους βοηθήσουμε. Κυρία Πρόεδρε, τι θα ήθελα να προτείνω εγώ να γνωστοποιήσουμε εμείς αυτό το πρόβλημα, να περαμείνει ανοιχτή αναφορά και θα είναι έτσι ευκαιρία για μια λεπτομερή μελέτη το τι συνέπειες έχει η κρίση σε αυτό το τομέα ναι μεν περισμένο σε μια ομάδα ατόμων, αλλά με τεράστια σημασία για να δούμε ακριβώς ε, τι είδους κοινωνία θέλουμε να οικοδομήσουμε στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μαρτίνες Μπάγκο. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ ότι είναι σωστά αυτά που λέει ο Αντιπρόεδρος Μαρτίνες Μαρτίν. Αλλά, αλλά, νομίζω ότι ο κύριος Μαρτίνεθ δεν είναι ενημερωμένος για την κατάσταση που επικρατεί στην Ουγγαρία και το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Εξάλλου, δεν μπορώ να εκτιμήσω την ακριβή κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο αναφέρον, αλλά το θέμα δεν είναι να ετοιμάσουμε άλλη μια μελέτη, είτε στην Ουγγαρία είτε αλλού. Η κυρία Κόντς ξέχασε να πει ότι τα τελευταία 15 με 20 χρόνια στην Ουγγαρία δημιουργήθηκε μια πραγματική βιομηχανία, ένας βιομηχανικός ο για τα επιδόματα ή τις συντάξεις για τους αναπήρους με πολλές απάτες. Αναπτύχθηκε επίσης ένα ολόκληρο σύστημα για να καταπολεμηθεί η κοινωνική αδικία. Γιατί πολλοί στα 40-45 τους χρόνια ε, ζητούσαν σύνταξη αναπηρίας, υποστηρίζοντας ότι είχα κάποια αναπηρία, και μετά συνέχιζαν να δουλεύουν παρά το γεγονός ότι παίρναν τη σύνταξη αναπηρίας. Η κυβέρνηση στην Ουγγαρία προσπαθεί να αντιμετωπίσει λοιπόν τέτοια φαινόμενα με ειδικού, με γιατρούς, με επιτροπές εμπειρογνωμόνων κλπ. Υπήρχε μία κατάσταση πολύ παραπημένη τελικά και από τις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες η Ουγγαρία ήταν αυτή η οποία είχε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό ανάπηρων από τις υπόλοιπες στην ίδια ηλικία. Στα 30, 40, 50 χρόνια έγινε σύγκριση και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι θέμα κράτους δικαίου, ούτε θέμα ε, νομικής ασφάλειας. Η Ουγγαρία είναι δημοκρατική χώρα που έχει τους θεσμούς που πρέπει να έχει. Η κυρία Γκόντς επίσης αναφέρθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Υπάρχουν όντως διάφορες προσφυγές που γίνονται στο ε, δικαστήριο, αλλά το δικαστήριο έχει απαντήσει. Ούτε η Επιτροπή Αναφορών, ούτε οι Ευρωβουλευτές έχουν δικαίωμα να ε, καταδικάζουν την κατάσταση στην Ουγγαρία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ξέρουμε ότι δεν περιορίζει το δικαίωμα των κρατών ε, μελών να καθορίζουν το δικό τους κοινωνικό σύστημα και κοινωνικών παροχών. Και εφόσον δεν υπάρχει νομοθεσία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι τα κράτη-μέλη αυτά τα οποία καθορίζουν τη δικιά τους νομοθεσία, βάσει της οποίας καθορίζονται οι προϋποθέσεις για να συνταξιοδοτείται κανείς ή να έχει κοινωνικές παροχές και ρυθμίζει βέβαια και τα ποσά. Από πλευράς κοινωνικής ασφάλισης, οι εξουσίε της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ περιορισμένες ακόμη και σε θέματα συντάξεων αναπηρικών. Συνεπώς, είναι σαφές ότι πρέπει να ζητήσουμε να κλείσει η αναφορά αυτή, διότι απλά δεν είναι κοινοτική αρμοδιότητα. Μπορεί να απευθυνθεί στα εθνικά δικαστήρια αναφέρον ή να πάει, αν έχει νομικό ζήτημα, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αλλά όχι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Γκόντς, για ένα λεπτό έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, λυπάμαι που επανέρχομαι. Λιγότερο από ένα λεπτό θα μιλήσω, αλλά θέλω να πω στον κύριο Μπάγκο, τον Ούγγρο συνάδελφο, ότι αυτά που λέει την Ουγγαρία δεν είναι ακριβώς έτσι. Κοιτάξτε, αυτές οι κοινωνικές ομάδες, οι πιο ευάλωτες που υποχρεωτικά εξαρτώνται από άλλους, υποφέρουν ακόμα περισσότερο από τις αλλαγές αυτές. Και σωστά λέτε ότι υπάρχουν διάφορες απάτες, διάφοροι που λένε ψέματα, σύμφωνα, αλλά υπάρχουν και πολλοί άλλοι οι οποίοι είναι πραγματικά ανάπηροι και όλοι υποφέρουν. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι συνταγματικές αλλαγές που γίνονται τώρα στη χώρα, το κόμμα που είναι στην κυβέρνηση προτείνει ακόμα να ε, θεωρείται έγκλημα η αναπηρία. Προσοχή, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Όπως είναι πάρα πολύ επικίνδυνο ξαφνικά ένας να έχει κάποιο δικαίωμα και ξαφνικά από τη μια μέρα στην άλλη να πάβει να το έχει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος. Θεωρώ ότι από τα όσα ακούσαμε στη συζήτηση επειδή είδαμε και την πλειοψηφία να εκφράζεται έτσι, δεν χρειάζεται να κλείσουμε αυτή την αναφορά, αλλά χρειάζεται απέναντι σε αυτούς τους πολίτες ε, να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από όσα είπε ο κύριος Μαρτίνες ε, η Επιτροπή να ερευνήσει τι σημαίνουν αυτές οι αυστηρές, οι μεγάλες περικοπές ε, στα διάφορα κράτη-μέλη και κατά πόσο περιορίζονται εγγυήσει σε δικαιώματα συνταξιοδότησης των πολιτών τους σε πολλές χώρες. Και η Επιτροπή δεν μπορεί να μας πει ότι δεν έχει αρμοδιότητες, αλλά σε πολλές χώρες επαναλαμβάνουμε όπως και στην Ιταλία, τη χώρα μου, σημειώθηκαν μεταρρυθμίσεις αλλαγές στο συντεξιωτικό σύστημα με νομοθεσίες ε, που έφεραν ε, τρομερά καταστροφικά αποτελέσματα. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός πολιτών, δεν ξέρω όμως ακριβώς, που δεν λαμβάνουν ακριβώς πια επιδόματα και λοιπά συντάξεις μετά από αυτή την υπό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσα συμφωνήθηκαν και με τον τρόπο που ρυθμίστηκαν. Άρα λοιπόν πριν να κλείσουμε την αναφορά θα πρέπει να καταβάλουμε αυτή την επιπλέον προσπάθεια. Θα ζητήσουμε με λεπτομεριακό σημείωμα να εξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλα αυτά που προέκυψαν από τη συζήτησή μας. Άρα λοιπόν παραμένει ανοιχτό το θέμα της αναφοράς αυτής. Στη συνέχεια η επόμενη αναφορά, η 10 του κυρίου Λορέντσο Τόρτο Ιταλικής Ιθαγένειας σχετικά με το δικαίωμα των ατόπων με αναπηρίες να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα. Ο κύριος Τόρτο έχει το λόγο για πέντε λεπτά. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Εγώ, Τόρτο Λορέντσο, υποφελούμε από την υπέροχη αυτή ευκαιρία να σας ευχαριστήσω όλους για την εξέταση της αναφοράς μου. Εγώ ταπεινά ο ίδιος ε, εδώ μέσα θα ήθελα να σας ε, παραθέσω ε, τα των αναπηρίες είναι πλούτος για τις χώρες μας ε, πολλά υποφέρουν τα άτομα με αναπηρίες και οι οικογένειές τους για να παραμένουν εγγυημένα τα δικαιώματά τους. Μέσα σε μια κοινωνία που δεν μας θεωρεί σαν ένα εθνικό πόρο πλούτο στο σύστημά τους, αλλά σε ένα βάρος ακριβώς επειδή δεν υπάρχει γνώση σε αρκετά άτομα του πώς έχει το θέμα και πολλά που δεν προσλαμβάνουν κόσμο με αναπηρίες. Στην Ιταλία ο νόμος 6899 είναι ένας νόμος που δεν υποχρεώνει όμως τον εργοδότη να προσλάβει κάποιον με αναπηρία σε περίοδους κρίσους. Ε, καταλαβαίνετε, μια εταιρεία που έχει δυσκολίες οικονομικές ε, δεν έχει πια αυτή, δεν αισθάνεται αυτήν την υποχρέωση να μας προσλάβει και ακόμα και άλλες εταιρείες ε, που δεν επιθυμούν άτομα με αναπηρίες πληρώνουν απλά και μόνο ένα πολύ χαμηλό πρόστιμο. Άρα λοιπόν λένε πληρώσαμε το πρόστιμο, δεν έχουμε πια καμία υποχρέωση να προσλάβουμε άτομα με αναπηρία και στην Ιταλία είμαστε περίπου 750.000 άτομα με φυσική αναπηρία που είμαστε στους καταλόγους ανεργίας και από αυτούς το 50 με 70% αναζήτησε εργασία, δεν πέτυχε κάτι και υπάρχει και ψηλότερο ποσοστό από αυτό το 50 σε 70% που βάσει στα στοιχεία του ΟΗΕ στις βιομηχανημένες χώρες δεν εργάζεται. Αυτό που μας απαντούν σχεδόν πάντα είναι, είναι το κλασικό θα σας πούμε αργότερα. Όλα αυτά είναι τρομερά και καταστροφικά. Η στρατηγική της Σαββόνας για την απασχόληση, την οικονομική ανάπτυξη που προωθείται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει το αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των ατόμων με αναπηρίες για μια ενεργή ένταξή τους στην κοινωνία, συμμετοχή τους στην κοινωνία και δυστυχώς οι άνεργοι διπλασιάστηκε ο αριθμός τους στην Ευρώπη σε σχέση με τα άτομα με τις συνήθεις ικανότητες. Και ακριβώς λυπάμαι γιατί η οδηγια 2078 δεν γίνεται σεβαστή που θα πρέπει να προβλέπονται από τους εργοδότες λογικές λύσεις για τα άτομα με αναπηρίες ώστε να μπορούμε και εμείς να εργαστούμε. Ο Ιταλικός νόμος αυτή την υποχρέωση δεν την προβλέπει απέναντι στους ε, εργοδότες και δεν υπάρχει αυτή η υποχρέωση απέναντι σε εκείνους που είναι άτομα με αναπηρία και επιτροπή στην αρχή του Απριλίου 2011 αποφάσισε να παραπέμψει το θέμα ε, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο γιατί ε, σημειώθηκε και μια σημαντική απώλεια, επαναλαμβάνω, θέσεων εργασίας για άτομα με αναπηρίες και βέβαια το θέμα αυτό το οποίο θίγω είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας ε, κάθε κράτος μέλους ξεχωριστά. Στην περίπτωσή μου της Ιταλίας. Αλλά θα ήθελα εδώ μπροστά σας ε, να φωνάξω μετά από όσα σημειώνονται σε όλη την Ευρώπη ότι έχουμε όχι μόνο τη θεσμική υποχρέωση αλλά και τη θυνηθική υποχρέωση να Περασπιστούμε τα δικαιώματα των ατόμων αναπηρία και των οικογενειών τους, γιατί αντιμετωπίζουμε την ε, αδιαφορία ή την αδικία την κοινωνική, γιατί ζούμε μέσα στον πόνο πολύ συχνά και καταλαβαίνετε ότι όποιος είναι σε ένα αναπηρικό καροτσάκι είναι δύσκολο να εξηγήσει τη θέση του. Σας ευχαριστώ για την προσοχή που μου αφιερώσατε. Σας ευχαριστώ. Η Επιτροπή έχει το λόγο. και πάλι στην κυρία Ιλάρια Μπρατσοντούρο. Στα Ιταλικά θα μιλήσω, λέει η ομιλήτρια. Η οδηγία αυτή καθορίζει το πλαίσιο για τη μάχη κατά της ε, διάκρισης και παίζει σημαντικό ρόλο για την ένταξη ατόμων με αναπηρίες ε, σε εργασία. Το άρθρο 5 αυτής της οδηγίας τι προβλέπει ειδικά οι εργοδότες στα άτομα με αναπηρίες να προσφέρουν λύσεις λογικές για να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση σε μια εργασία, να μπορέσουν να ασχοληθούν και να μπορέσουν και να προχωρήσουν στη σταδιοδρομία τους. Και εμείς στην άσκηση των καθηκών μας ξεκινήσαμε μια προσφυγή επί παραβάση κατά της Ιταλίας, γιατί κατά την άποψη της Επιτροπής μας δεν εφαρμόζει όπως πρέπει το άρθρο 5 της οδηγίας αυτό έγινε τις αρχές Απριλίου του 2011 προσφύγαμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, προωθείται η διαδικασία και ακριβώς σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβιάζει το άρθρο 5, τότε θα πρέπει στην οδηγία 2078 να προσαρμοστεί η Ιταλική νομοθεσία. Το άρθρο 7 της οδηγίας επιτρέπει στα κράτη-μέλη να διατηρεί ή να υφετεί ειδικά μέτρα για να αντισταθμίσει τα όσα ε, αρνητικά συμβαίνουν λόγω αναπηρίας κάποιου ατόμου. Η οδηγία 2078 δεν προβλέπει όμως μια ειδική υποχρέωση για τα κράτη-μέλη, δηλαδή από διαφορετικής πλευράς ε, να απαλείψει τις διαφορές, όπως αναφέρεται εδώ στην αναφορά. Η πολιτική δημιουργίες θέσεων εργασίας και για άτομα αναπηρία είναι αποξηγής αρμοδιότητας των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν αναγνωρίζει βέβαια τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν άτομα με αναπηρία στην Ιταλία, αλλά διαπιστώνει ότι όλα αυτά που αναφέρονται ακριβώς ε, αρμοδιότητες αποκλειστικής επαναλαμβάνουμε του κράτους μέλους, δηλαδή στην περίπτωση αυτή της Ιταλίας. Κάποιος άλλος θα επιθυμούσε το λόγο, λέει η Πρόεδρος Μαρτίνες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως αντιλαμβάνεστε και θα συμβαίνει και με άλλους που μας νοιάζει η αλληλεγγύη, ε, είναι να, να όταν ακούς αυτά που λέω αναφέρον. Ραγίζει η καρδιά σου. Σίγουρα πρέπει να προχωρήσουμε. Οπότε, ε, με εκπλήσει κάτι από αυτά που ακούω. Σε ένα θέμα τόσο ξεκάθαρο. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει δύο χρόνια χωρίς να καταλήξει σε απόφαση. Ε, δεν ξέρω η δικιά μας Επιτροπή τι μπορεί να κάνει για να κάνει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να προχωρήσει. Είναι παράδεκτο αυτό. Και για ένα θέμα το οποίο δεν χρειάζεται στο κάτω-κάτω καμιά μεγάλη έρευνα από την ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο αναφέρον. Είναι ένα θέμα που είναι ξεκάθαρο ότι η Ιταλία δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της. Γιατί δεν έχει ενσωματώσει αυτή την οδηγία. Συνεπώς, πέρα από το ότι πρέπει να απευθυνθούμε στις Ιταλικές αρχές, θα ήταν καλό η πρόεδρός μας να στείλει μία επιστολή όπου να εκφράζει τη δυσαρέσκεια της Επιτροπής μας αλλά και την έκπληξή μας για το γεγονός ότι δεν έχει προχωρήσει. Το δικαστήριο θέλει δύο χρόνια για να καταλήξει σε απόφαση για αυτό το θέμα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Α, ίσως ναι, κάτι ακόμα. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και είναι καλό να το ξέρει αυτό ο αγαπητός Τόρτο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν φροντίζουμε να τηρούμε τους κανόνες για να προσλαμβάνουμε άτομα με αναπηρίες. Και σε πολλούς τομείς εργασίας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθημερινά διαπιστώνουμε ότι έχουμε συναδέρφους με κάποια αναπηρία. Και να είσαστε σίγουροι ότι η δουλειά που προσφέρουν είναι πάρα πολύ ικανοποιητική. Απόλυτα ικανοποιητική. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λοιπόν, μπορεί να μην το γνωρίζουν όλοι οι συνάδελφοι, αλλά εμείς που το γνωρίζουμε, το διαπιστώνουμε καθημερινά και εμείς που γνωρίζουμε κάποια από αυτά τα άτομα με αναπηρίες, είμαστε, πρέπει να ξέρετε, απόλυτα ικανοποιημένοι από το έργο τους. Διαπιστώνουμε δηλαδή καθημερινά ότι δεν κάναμε λάθος που εφαρμόσαμε αυτούς τους κανόνες για την πρόσληψη ατόμων με αναπηρίες. Τα άτομα αυτά φέρουν σε πέρα στην εργασία τους χωρίς κανένα πρόβλημα, απόλυτα ικανοποιητικά. Γι' αυτό κυρία Πρόεδρε νομίζω ότι θα ήταν καλό να ε, στείλουμε επιστολή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ζητώντα του να δραστηριοποιηθεί για αυτό το θέμα και να προχωρήσει σε απόφαση, μια που μας μοιάζει πάρα πολύ. Ο κύριος Γιάρ. Να συμπληρώσω κι εγώ αυτό που λέει ο συνάδελφος. Να ζητήσω κι εγώ η Κομισιόν να προειδοποιήσει την Ιταλία να εφαρμόσει την τη 2078 γιατί όταν διαβάζουμε το κείμενο λέει ότι σύμφωνα με αυτή την οδηγία ο, εργαζ... ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος σύμφωνα με να ε, λάβει κάποιες πρόνοιες για τα άτομα με αναπηρία για να τους εγγυηθεί την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας. Η Κομισιόν, λοιπόν, λέει ότι δεν έχει εφαρμόσει πλήρω η Ιταλία την οδηγία αυτή. Για μένα λοιπόν ισχύει αυτό που ζητά ο αναφέρον. Φυσικά πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις διαρθρωτικές, τα διαρθρωτικά προβλήματα που μπορεί να έχουν τα κρατημέλη, αλλά το αίτημα καλύπτεται ουσιαστικά, δεν καλύπτεται από το ότι δεν, ε, δεν εφαρμόζεται αυτή η οδηγία. Οπότε η Κομισιόν πρέπει να προειδοποιήσει την Ιταλία ότι πρέπει να ε, την εφαρμόσει την οδηγία 2078. Ίσως ε, να μην, ε, ε, να μην αξίζει να καθυστερήσουμε εδώ για λόγους τακτικής. Το θέμα είναι ότι εδώ μιλούμε για ανθρώπους αδύναμους, τους πιο αδύναμους της κοινωνίας και πρέπει μέσω της Κομισιόν ή η Ιταλία να υποχρεωθεί επιτέλους να εφαρμόσει την οδηγία. Ευχαριστώ. Ο αναφέρον έχει το λόγο για να απαντήσει. Σας ευχαριστώ όλους. Εκ βάθους καρδίας εύχομαι ότι όποιος υποφέρει όπως εγώ και πολλοί άλλοι που ζουν μέσα στη σιωπή γιατί δυστυχώς υπάρχουν και άτομα που δεν μπορούν να εκφραστούν ε, όπως εγώ σήμερα που είμαι εδώ, έχω την τύχη να βρίσκομαι εδώ και να σας διηγηθώ μια τρομερή πραγματικότητα. Αυτή η ταπεινή φωνή μου θέλει να βοηθήσει και πάρα πολύ κόσμο που δεν τα καταφέρνει και πολλές οικογένειες που παραμένουν μόνες και αυτό για το κράτος μέλος. Το κράτος μέλος δεν έκανε το καθήκον του. Γι' αυτό σας παρακαλώ να είσαστε εσείς οι φύλακες, οι προστάτες. Όχι για μένα, είμαι μικρός και ταπεινός, αλλά για πάρα πολύ κόσμο που χρειάζεται τη βοήθειά σας. Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε την κατάσταση. Γιατί για κάποιον που υποφέρει ο χρόνος είναι τύρανος. Όποιος έχει προβλήματα παρόμοια δεν μπορεί να περιμένει έτσι τα όσα ισχύουν θεσμικά, διαδικαστικά κλπ. Και μια δικαιοσύνη που αργεί να εφαρμοστεί. Και όταν αργεί να εφαρμοστεί, κυρίως για τους ασθενέστερους, ξέρετε τι σημαίνει. Είναι μια αδικία μεγάλη. Κάποιος ε, που έχει προβλήματα αναπηρίας καταδικάζεται δύο φορές και γιατί υποφέρει από την αναπηρία του αλλά επειδή δεν μπορούμε να σου προσφέρουμε και μια καλύτερη ζωή και επειδή είναι σύντομη η ζωή πρέπει να και θέλω να ελπίζω ότι κάτι το θετικό κάνω. Γι' αυτό να προσθέσω, επαναλαμβάνω τα ταπεινά μου λόγια για να βοηθήσω ώστε να αλλάξω όχι την ιστορία, δύσκολο, δεν αλλάζει, αλλά η ιστορία αλλάζει σιγά σιγά με μικρές κινήσεις. Αλλά τουλάχιστον να δώσουμε να καταλάβουμε, να καταλάβουν αυτά τα άτομα ότι πρέπει να βοηθηθούν, μπορούν να βοηθηθούν και όταν δεν μπορεί κάτι να κάνει το κράτος να τα πείτε εσείς. Κάποιος ε, πάτερ φαμίλιας που θα πει στην οικογένειά του «Ε, εσύ δεν είσαι πια σωστός, πρέπει να με ακούσεις. Εδώ είστε μια μεγάλη οικογένεια, η Ευρώπη για όλους μας θα πρέπει να είναι μια μεγάλη οικογένεια θεματοφύλακας όλων αυτών των αξιών που θα πρέπει να μας διακρίνουν παντού και πάντα πρέπει να είναι ο οίκος εκείνου που υποφέρει. Όχι γιατί υποφέρω εγώ προσωπικά, ατομικά, γιατί υποφέρουν πολλοί. Θα πρέπει να δείξει τη δύναμή σας για όλους. Σας ευχαριστώ από βάθους καρδιάς και καθένα ένα ξεχωριστά, γιατί μου δώσατε αυτή τη δυνατότητα. Όχι, όχι, δεν είστε ένας φορέας φιλανθρωπίας, αλλά να σας πω ότι χαίρομαι που ήρθα εδώ. Χαίρομαι που μπορούσα να τα πω αυτά. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ όλοι πρόεδρος. Ευχαριστούμε τον κύριο Τόρτο. Ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας και εγώ η ίδια σαν Ιταλίδα υπήκος εκφράζω την απογοήτευσή μου για όσα συμβαίνουν. Το γνωρίζω τα πράγματα και σαν εθνική βουλευτής πολλές φορές με δικές μου νομοθετικές πρωτοβουλίες προσπάθησα να αλλάξω μια κατάσταση που θεωρώ εντελώ απαράδεκτη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, προσπάθησε να αλλάξει την κατάσταση ήδη το 2006 με μια προσφυγή επί παραλήψη ακριβώς επειδή δεν σεβάθηκε η Ιταλία την οδηγία αλλά τώρα μπροστά σε αυτό το ευρωπαϊκό επίπεδο να δούμε πως μια προσφυγή επί παραλήψη τι γίνεται το 2006 κατατέθηκε αλλά το 2013 παραμένει σε κρεμότητα δεν είναι άσχημα τα πράγματα, δεν είναι η κατάσταση, τρομερή κατάσταση. Μετά από τόσα χρόνια δεν καταφέραμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα. Γιατί όπως το είπατε ο ίδιος, σε παρόμοιες καταστάσεις, σε παρόμοιες δυσκολίες έχει ιδιαίτερη σημασία ο χρόνος και το πέρασμά του. Άρα λοιπόν όπως είπαν και ορισμένοι συνάδελφοι, θα απευθυνθούμε και στο δικαστήριο και θα του ζητήσουμε μια επιτάχυση της όλης ε, διαδικασίες και θα ζητήσουμε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιταχύνει και εκείνη το ρυθμό της για όλες τις προσφυγές επί παραλήψη, γιατί απλά και μόνο μια απειλή δεν ωφελεί σε τίποτα από τη στιγμή που περνάνε τόσα χρόνια και μπορεί να συνεχίσει το κράτος αυτό να ενεργεί χωρίς να σέβεται τις υποχρεώσεις του γιατί προσφυγή επί παραλήψη σημαίνει ότι δεν σεβάστηκαν υποχρεώσεις τους και δεν μπορεί να το παραγνωρίζει αυτό το γεγονός η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά και σας ευχαριστώ. Κλείνουμε με το σημείο αυτό της ημερήσιας διάταξης. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, το θέμα του κυρίου Μακμίλαν Σκότ. Πρόκειται για μια πρώτη εξέταση για τις δραστηριότητες της Επιτροπής μας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι που μπορώ να σας παρουσιάσω το σχέδιο του εξηγηματικού σημειώματος ε, για τις δραστηριότητες ε, της Επιτροπής ε, Αναφορών 2012. Η Επιτροπή αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική. Δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ακούσαμε από τους αναφέροντες σήμερα το πρωί. Μα επιτρέπει επίση να παρακολουθούμε την εφαρμογή των, ε, της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας από τα κράτη-μέλη σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, τη κράτη-μέλη και την Κομισιόν αλλά και την Κοινωνία των Πολιτών. Περιμένουμε βέβαια στα στατιστικά στοιχεία. Θα δείτε ε, πολλά ε, σημεία που είναι κρεμή στην, ε, στο σχέδιο, όπως είναι η προστασία των δικαιωμάτων, η ιστορική αγορά, η υγεία και η ευζοία των ζώων. Ε, χαίρομαι που μπορώ να πω ότι ήταν επιτυχής ο χρόνο αυτό για την Επιτροπή. Δεν θα σα αναφέρω όλε τι ε, λεπτομέρειες. Θα επικεντρωθώ μόνο σε κάποια σημεία. Μία θετική εξέλιξη τη δουλειά μα ήταν ε, η δημιουργία τη άτυπη ομάδα εργασία για τα ε, δικαιώματα ιδιοκτησία στην Ισπανία. Ξέρετε ότι από το 1984 βρίσκομαι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχω κάνει πολλέ αναφορέ για το θέμα αυτό, κυρίω για την Ισπανία και την Πορτογαλία, όταν πρόκειται να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έτσι καταλήξαμε σε μια έκθεση του 1988 σχετική. Ε, έχουμε συναντηθεί με, υπουργο... με εκπροσώπους των Ισπανικών Υπουργείων. Υπάρχει μια συνάντηση στην Ισπανία αύριο που θα γίνει και οι συνάδελφοι έχουν λάβει ήδη τον σχετικό φάκελο από την Γραμματεία. Αυτό ο τελευταίος χρόνο επίσης έδειξε ε, πόσο σωστή είναι η ε, ε, πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών όπου μπορούμε να έχουμε ανεξάρτητη οργάνωση διαφόρων ακροάσεων μαζί με την συνήθη δουλειά που κάνουμε. Η έκθεση για το 2011 από τον συνάδελφο Τσίτσεστερ δείχνει ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα αποτελούν, τα, αποτελούν το αντικείμενο κατά μεγάλο βαθμό των διαφόρων αναφορών και η, η, Λίμπε έχει κάνει μια σχετική ε, έκθεση από τη συνάδελφο Βάλιαν όπου αναφέρεται ότι ε, ε, η διακριτική μεταχείριση δεν θα πρέπει να γίνεται με βάση τις θρησκευτικές πεπιθήσεις, τις πολιτικές πεπιθήσεις, το φύλλο το κτλ. Επίσης, είχαμε τη θέση μας για, το, για την άκτα με σε εσάς κυρία Πρόεδρε και με τον David Martin που ήταν ο εισηγητής και που έλαβε την ε, ε, αναφορά με περίπου 2,5 εκατομμύρια ε, υπογραφές που ήταν αντίθετες με την άκτα λόγω του ότι παραβιάζει θεμελιώδεις ελευθερίες. Μετά το 2000, τον Ιούνιο του 2012 η αντίθεσή μας στην άκτα οδήγησε στην αρνητική ψήφο του Κοινοβουλίου επ' αυτού. Το έγγραφο εργασία για την διαρνητική επίσκεψη στο Βερολίνο επίση υιοθετήθηκε, τονίζοντα τι τις ε, ε, πρακτικές διακριτικής μεταχείρισης ε, κάποιων οργανώσεων που ασχολούνται με την προστασία παιδιών. Υπάρχουν βεβαίω εκκρεμή θέματα σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των παιδιών που πρέπει να κλείσουν και πιστεύω ότι αυτά θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην έκθεσή μου. Η ηθαγένεια επίση είναι ένα σημαντικό κομμάτι τη έκθεση. Το 2012 αποφασίσαμε ότι το 2013 θα είναι το έτο του πολίτη και έχουμε μία ε, έκθεση πρωτοβουλία από το 2010 από την κυρία Βαλιάν πάλι, η οποία έχει οθετηθεί. Ε, επίσης, μελετήσαμε την, ε, τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης στην Ιθαγένεια με συγκεκριμένο πλάνο που θα διεξαχθεί φέτος. Το παρεβάλλον επίσης είναι σημαντικό τομέα της έκθεσης. Το σημείο μα μιλάει για τη διάθεση αποβλήτων. Επίσης υπάρχουν αναφορές που μας ευστούν την προσοχή στις αρνητικές συνέπειες ε, διαφόρων πρακτικών ε, εξόρυξης ε, και άλλων. Πράγματα που συμβαίνουν και στη δική μου την εκλογική περιφέρεια του Yorkshire. Επίσης θα παρουσιάσω μια, ένα σχέδιο έκθεσης στις 24 Απριλίου με συγκεκριμένα στατιστικά δεδομένα. ελπίζω ότι θα, έχουν, θα υπάρξουν ανθρωπολογίες μέχρι τον Μάιο και θα γίνει ψηφοφορία στην Επιτροπή τον Ιούνιο και το Σεπτέμβρη θα, γίνει, θα τεθεί σε ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο. Αυτό το σχέδιο είναι ακόμα εν εξελίξη και βεβαίω καλωσορίζω τα σχόλιά σα. Ένα τελικό σχόλιο είναι ότι πρέπει να, ε, ευχαριστήσω την Πρόεδρο γιατί έλαβε την ε, σύμφωνη γνώμη του Πρόεδρου Σούλτς ώστε η Επιτροπή να μελετήσει ε, τους ε, αναφέροντες, ε, τους μεμονωμένους αναφέροντες που έρχονται στις Βρυξέλλες είναι περίπου 1.700.000. Ε, Το έχει αναλάβει ο κύριος Τσίσεστερ και η ΑΦΚΟ κάνει μια σχετική συζήτηση για τη δική της σχετική έκθεση. Μάλλον την έκανε χτες. Και τέλος να ευχαριστήσω τους υπαλλήλους της Επιτροπής που βοήθησαν για την σύνταξη αυτής της, αυτού του σχεδίου και ελπίζω ότι η δουλειά μας θα είναι εξίσου αποδοτική και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και μάλιστα διπλά συνάδελφε Μακμίνταν Σκοτ κυρία Τζανοκά Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Μακμίλαν Σκοτ Η δουλειά σας συνοψίζει πολύ καλά το δικό μας έργο κατά τη διάρκεια του 2012 Η ερώτησή μου είναι η εξής. Μπορεί να ασφάλω, κύριε Ντέιβιτ Λό, αλλά δεν έχουμε και την έκθεση για την επίσκεψη στο Γιόρτζορ το 2012, δεν έγινε, που επίσης είχε να κάνει με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα δικαιώματα των οικογενειών και την χρήση της γλώσσας. Ξέρετε όλες αυτές τις ε, αναφορές που είχαν να κάνουν με την απαγόρευση των παιδιών να μιλούν ε, τη γλώσσα τους. Και το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει επειδή οι οικογένειες πολλές φορές αναγκάζονται να ζουν χωριστά και δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την γλώσσα τους. Υπάρχει διάκριση δηλαδή επειδή ανήκουν σε μία γλωσσική μειονότητα. Άρα είναι παραβίαση της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Θα ήθελα λοιπόν να το υπενθυμίσετε και αυτό, να συμπεριλαμβάνετε και αυτό στην έκθεση υπεπραγμένων για το 2012. Παρακαλώ, κύριος Κάσης. Ναι, ευχαριστώ, ευχαριστώ πρόεδρε. Συγχαρτήρια στον κύριο Μακλήραν Σκότ για την εργασία του αυτή. προκαταρτική εργασία είναι αυτή και εδώ για την Επιτροπή Αναφορών φαίνεται το εύρος της ευθύνης ε, μας για την υπεράσπιση των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη συζήτηση αυτή η σχέση ανάμεσα στην ευρωπαϊκή ηθαγένεια και στο δικαίωμα αναφοράς είναι κάτι με ιδιαίτερα μεγάλη σημασία. 2012-2013 είναι σημαντικά δύο χρόνια για την ευρωπαϊκή ηθαγένεια και για τους καταναλωτές σαν πολίτες οι ίδιοι. Και θα πρέπει να συντάξουμε την έκθεση αυτή και σωστά και έχει μεγάλη σημασία. Αυτή η ευρωπαϊκή ηθαγένεια αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο και θα πρέπει να αποκτήσει σώμα και στο μέλλον θα είναι από τους ε, σημαντικούς τρόπους ε, πραγματοποίησης και υπεράσπισης αυτής της ιθαγένειας στα θεσμικά μας όργανα. Γι' αυτό ακριβώς δεν θα πρέπει όμως να ξεχνάμε και την οικονομική και κοινωνική κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το τι προκαλεί, όπως το είπαμε ήδη. Για τα θεμελιώδη δικαιώματα, δικαιώματα πραγματικά κλειδιά που έχουμε πετύχει αυτά τα τελευταία χρόνια και είδαμε ας πούμε με τα περισσότερα ευάλωτα άτομα να υποφέρουν όπως και τα άτομα με αναπηρίες. Έχει σημασία επίσης ε, εδώ στην Επιτροπή μας και με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου να δείξουμε ποια είναι η θέση μας με την ε, ελευθερία έκφρασης ε, την δοτική σφαίρα και την δυνατότητα δράσης και ενέργειας του καθένα μας. Και εδώ για το 2012 θυμάμαι τη θέση που έχουμε υιοθετήσει για όσους έχουν εκτελεστεί την ε, περίοδο του Φράνκο στην Ισπανία και πώς θα έχει πρόσβαση κανείς σε στοιχεία να δει πώς συνέβησαν, κατά ποιες συνθήκες συνέβησαν όλα αυτά. Και είναι επίσης το θέμα των ε, απαχθέντων ε, παιδιών ε, από το 1940 μέχρι το 1990 στην Ισπανία. και επίσης να υπερσπιστούμε το περιβάλλον, την δημόσια υγεία, όλα αυτά με σημαντικό μέρος του στο 2012 και στο μέλλον βέβαια αποτελεί ένα σημείο πάντα σημαντικό και θα είναι ακόμα πιο σημαντικό επίσης για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και το πώς επηρεάζουν την υγεία όπως επίσης να δώσουμε προτεραιότητα στην πρόληψη μπροστά σε όλη αυτή την εξέλιξη της βιοτεχνολογίας. Κάτι το τελευταίο και εδώ ολοκληρώνω. Δείξαμε ιδιαίτερη ευαισθησία και διατηρούμε τις θέσεις μας για τα ύδατα, ότι είναι κοινό αγαθό. Όπως επίσης και εδώ σε διάφορες στιγμές το έχουμε υπερασπιστεί αυτό για τη χρήση, τη διαχείριση των υδάτων ε, πρέπει να είναι από τα σημαντικά στοιχεία για τους Ευρωπαίους πολίτες τα χρόνια που θα ακολουθήσουν αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε. Ο... Η κυρία Βάσκο ζήτησε το λόγο. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ως ε, σκιώδης ε, του ΕΛΚ ε, θέλω και εγώ να αναφερθώ στα πεπραγμένα μας για το 2012. Η έκθεση αυτή έχει ως στόχο να δείξει στους πολίτες ότι τους εκπροσωπούμε σωστά σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ότι όλες οι αναφορές τους τυχαίνουν καλή μεταχείρισης εδώ, ότι τις ασχολούμαστε, τις επεξεργαζόμαστε όπως τους πρέπει. Έχει πολύ μεγάλη σημασία βέβαια η πληροφορία που μας δίνουν οι πολίτες που Δυστυχώς βάσει του ευρωβαρομέτρου βλέπουμε ότι οι πληροφορίες που φτάνουν από εμά τους πολίτες δεν είναι αρκετές. Μόνο 25% των πολιτών λένε ότι υποφελούνται από τις πληροφορίες αυτές. Ούτε μπορούν να κάνουν διάκριση ανάμεσα στα διάφορα θεσμικά όργανα. Μερικές φορές τις αναφορές τους δεν τις θέλουν καν στο σωστό όργανο. Η έκθεσή μας επίσης βασίζεται σε διάφορα στατιστικά δεδομένα. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει κεντρική διάθεσή τους. Για παράδειγμα, ποιες είναι οι αναφορές που έχουν καταγραφεί, ποιες έχουν δεχτεί οι παραδεκτές, ποιες έχουν κλείσει και ποιοι είναι οι τομείς αναεθνικότητα που, ε, των αναφορών που φτάνουν σε εμά. Πρέπει να Συζητήσουμε λοιπόν για την έκθεση αυτή, διότι έχουμε 60 αναφορές που δεν έχει αποφασιστεί το κατά πόσο είναι παραδεκτές ή όχι. Το 2012 οι περισσότερες αναφορές που υποβλήθηκαν είχαν να κάνουν με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Εδώ θα πρέπει να επενθυμίσουμε ότι υπάρχει αποκλεισμός των Αθήγανων, των Ρώμα, κάτι το οποίο τους βάζει σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Και πάνω πολλά χρόνια που έχει ξεκινήσει η σχετική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ένταξη των ατόμων αυτών. Πρέπει επίσης να προετοιμαστούμε για το 2013 και να προβλέψουμε μία έκθεση για τα στατιστικά δεδομένα και για τα πιο σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα την προηγούμενη χρονιά. Η ομάδα εργασίας, ε, για παράδειγμα, που δημιουργήθηκε για το αέριο σχιστόλιθου όπου έγιναν συζητήσεις ανοιχτές και πολύ ενδιαφέρουσες στην Επιτροπή μας. Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα είναι οι δραστηριότητες της Επιτροπής μας για το 2012, ε, μεταξύ άλλων οι επισκέψεις μας στην Ιταλία στα τέλη Οκτωβρίου. Με αυτόν τον τρόπο, με τις επισκέψεις αυτές, μπορούν επιτόπου να δουν οι προβουλευτές τι έγινε με τα απολύματα στο Λάτσιο και στην Καπάνια. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό που αξίζει τον κόπο να αναφέρουμε είναι η θέση σε ισχύ από την 1η Απριλίου του 2012 της πρωτοβουλίας των Ευρωπαίων πολιτών. Μια πρωτοβουλία η οποία αποτελεί μια μοναδική περίπτωση δυνατότητας έκφρασης των Ευρωπαίων πολιτών, οι οποίοι έτσι μπορούν πολύ δραστήρια να συμμετάσχουν στις αποφάσεις μας. Πιστεύω ότι η έκθεση αυτή πρέπει να επενθυμίζει και την εξαίρετη συνεργασία που έχουμε με τον ε, Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Αυτά λοιπόν είναι τα κύρια θέματα που είχα να αναφέρω και ελπίζω να έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με τον εισηγητή αλλά και τους άλλους σκιώδεις εισηγητέ. Τώρα, αν άλλοι ευρωβουλευτές έχουν προτάσεις όσον αφορά το περιεχόμενο της έκθεσης αυτής για το μέλλον, θα πρέπει να τις λάβουμε υπόψη μας. Υπενθυμίζω επίσης ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η Δευτέρα Μαΐου. 2 Μαΐου προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, κύριε Μακμίλαν ε, Σκοτ, και πάλι έχετε εσείς το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Άκουσα τα σχόλια της κυρίας νόκα. Όντως, η περίπτωση της επίσκεψης αυτής ε, είναι κάτι σημαντικό. Τώρα οι προσπάθειες της Επιτροπής μας αλλά και άλλων επιτροπών για αλλαγές για να συμπεριληφθεί ας πούμε η χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων, τα δικαιώματα των παιδιών, να προσθέτει και τα δικαιώματα των γονέων. Υπάρχει μια συνάντηση αυτή την εβδομάδα στο γραφείο μου με πατέρες, με οργανώσεις δηλαδή που εκπροσωπούν ε, πατέρες παιδιών που έχουν ε, απαχθεί που δεν μπορούν να τα δουν. Είναι ένα θέμα όντως πολύ σημαντικό. Ο κύριος Γκάθια πολύ σωστά από την άλλη υπογράμμισε τη σημασία που έχει η οικονομική κρίση. Όπως είπα και στην αρχή, θα έχουμε ακρόαση, αλλά υπάρχουν πολλά ζητήματα που έθεσαν το 2012 οι αναφέροντες και που έχουν να κάνουν με την οικονομική κρίση, πράγματι. Η κυρία Παντέσκου είναι σκιώδης από το ΕΛΚ, πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Εννοείται ότι και εγώ προσβλέπω σε στενή συνεργασία μαζί της και με τους άλλους σκιώδης εισηγητές. Πολύ σωστά λέει ότι η έκθεση αναφέρει τις πιο σημαντικές περιπτώσεις, δραστηριότητες ή αναφορές της χρονιάς που πέρασε. Αντιλαμβάνομαι ότι πέρυσι ήταν κάπως δύσκολη κατάσταση υπήρχε πίεση προς διαφορετικές κατευθύνσεις και έπρεπε να καταλήξουμε σε μια ισορροπία. Εγώ χρησιμοποιώ την δικιά μου μακρά εμπειρία στο χώρο για να συντάξω την έκθεση αυτή. Κατά τα άλλα είμαι ανοιχτό. Όμως η έκθεση πρέπει να αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή μας πέτυχε πολλά και μην ξεχνάμε ότι θα είναι και η τελευταία πριν από τι ευρωεκλογέ. Γι' αυτό και πρέπει να αντικατοπτρίζει πάρα πολύ καλά τι προσπάθειε που έχουν κάνει διάφοροι ευρωβουλευτέ μέλη τη επιτροπή αυτή. Γιατί περί αυτού πρόκειται στι εκλογέ. Γι' αυτό και θέλω να επικεντρωθώ πάρα πολύ στου ευρωβουλευτέ που προσέφεραν αξιόλογο έργο στην Επιτροπή αυτό και βοήθησαν να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Αυτά, τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Σα ευχαριστούμε κύριε Μακμίλαν Σκοτ. Εντάξει, θα προχωρήσουμε και με όσα λέτε τώρα, μετά από όσα ακούσατε. Τελειώνει η εργασία μας για σήμερα το πρωί. Λίγα λεπτά διάλειμμα, παύση για να συνεχίσουμε με τους συντονιστές. Σας ευχαριστώ όλους.